Okay, um, Συνάδελφοι, ξεκινήσουμε. Λυπάμαι που ήμουν απούσα σήμερα το πρωί. Άφησα στην κυρία Τρούπελ όλη τη δουλειά. Ήμουνα στο Βερολίνο εχθές για, την εορτασμό, για τον εορτασμό των, ε, ε, των 50 χρόνων της συνθήκης των Ελυσίων ε, και επειδή είμαι δίπλα στα γαλλικά σύνορα, έπρεπε να πάω και στη Γαλλία για να γιορτάσουμε και από εκεί. Σήμερα το πρωί έκανα και μια ομιλία για τον ε, πολιτισμό και για τον εορτασμό βεβαίως των 50 χρόνων της συνθήκης. Χαίρομαι που τελικά έφτασα εδώ και είναι και η κατάλληλη στιγμή, γιατί έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς προστεκλημένους. Έχουμε εκπροσώπους των ε, της Ιρλανδικής Προεδρίας, οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα να λύσουν. Έχουμε το νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, το νέο πρόγραμμα για, την, για τον πολιτισμό, το πρόγραμμα για την Ευρώπη των πολιτών και έχουμε και την πολιτισμική πρωτεύουσα. Ένα μεγάλο πακέτο λοιπόν, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της δικής σας Προεδρίας και τώρα θα περάσω στα γερμανικά. Ε, τώρα αφού έχουμε τους αγγλόφωνους εδώ, ας μην ε, ε, παρουσιάσω εγώ το, τα κακά μου αγγλικά. Λοιπόν, χαίρομαι που είσαστε σήμερα εδώ τις, ε, τους τελευταίους μήνες έχουμε κάνει πολλή δουλειά στην Επιτροπή μας, έτσι ώστε να υπάρξει συμπλήρωση, βελτίωση, ενίσχυση των όσων έχει προτείνει η Κομισιόν, για να μπορέσουμε από κοινού με να προχωρήσουμε για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Αν δεν τα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα στην δική σας Προεδρία, θα έχουμε δυσκολίες να ε, μπορέσουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα αυτό το 2014. Γι' αυτό σας έχουμε εμπιστοσύνη και Ξέρουμε ότι σε κάποιους τομείς υπάρχει μια μερική γενική θέση. Ευτυχώς δεν είναι το τέλος αυτό. Είναι όμως μια θέση που είναι διαπραγματεύσιμη και εμείς έχουμε τη διάθεση να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και των ψηφοφοριών μας Χωρί όμω να ε, επιδεινώσουμε την ε, φιλικότητα προ το χρήστη όλων αυτών των ε, προγραμμάτων και βεβαίω έχοντα υπόψη ότι όλα αυτά που ζητούμε πρέπει με κάποιο τρόπο να βρίσκονται μέσα στο πρόγραμμα. Θα μιλήσουμε για πρώτη φορά για το πρόγραμμα για τον αθλητισμό, για τον αθλητισμό το οποίο όμω μπαίνει στο γενικότερο πλαίσιο του πρόγραμματο για την εκπαίδευση και χαίρομαι που σήμερα έχουμε δύο υπουργού εδώ. Ο τρίτο, δυστυχώ για οικογενειακού λόγου δεν μπόρεσε να είναι μαζί μα. Έχουμε λοιπόν εδώ μαζί μας τον Υπουργό Πολιτισμού, ο κύριος Κάνον, όχι. Συγγνώμη, ο κύριος Ρίνκ και ο κύριος Ντένιχαν είναι μαζί μας σήμερα. Ωραία, πολύ ωραία. Ε, έχουμε λοιπόν τον κύριο, ε, τον Υπουργό Ντένιχαν, Υπουργό τεχνών κληρονομιάς και γαλλικών υποθέσεων. Ωραία ακούγεται αυτό το γαλλικών υποθέσεων. Πολύ ωραία. Και έχουμε και τον Υπουργό Ρίνγκ ε, να αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμό, ο οποίος θα μας μιλήσει αργότερα. Πρώτα, ο Υπουργό Τένιχαν έχει το λόγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Πακ για την Επιτροπή σας για την ευκαιρία να παρουσιάσω τις βασικές προτεραιότητες της Ιρλανδίας για τον πολιτισμό κατά τη διάρκεια της Θέλω να παρουσιάσω και τους συναδέλφους μου, ο κύριος Ρεν, υπουργό και δύο αξιωματούχοι, ο κύριος Τέλη από το, το γραφείο μου στο Δουβλίνο. Θέλω να ξεκινήσω τις παρατηρήσεις μου λέγοντας ότι οι τέχνες ήταν πάντα ένα στο τμήμα της Ιρλανδικής ζωής και ότι μέσω του Culture Connect, το, προ, το πρόγραμμα της προεδρίας μας, θέλουμε να δείξουμε τη δύναμη της ποικιλομορφίας της κουλτούρας στην Ιρλανδία και στην Ευρώπη και να υπογραμμίσουμε την κοινή φύση πολλών από τις πολιτισμικές μας εμπειρίες. Το πρόγραμμα θα επιδιώξει να κάνει κάτι τέτοιο με την εμπλοκή Ιρλανδών καλλιτεχνών στην πατρίδα μας, στην Ευρώπη και πέραν της Ευρώπης, παρέχοντας δυνατότητα σε Ευρωπαίους καλλιτέχνες να έρθουν στην Ιρλανδία και να δουλέψουν δημιουργικά μαζί για να εμπλουτίσουν τις σκέψεις μας στην Ευρώπη και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013, τα 40 χρόνια της προσχώρησής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1973. Η ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών με σεβασμό της πολιτισμικής διαφορετικότητας και την ενίσχυση του οικονομικού ρόλου του πολιτισμού και των δημιουργικών τομέων πρέπει να είναι στο κέντρο αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε στον πολιτισμικό τομέα τα επόμενα έτη. Η βασική προτεραιότητα της Ιρλανδίας είναι να σταθούμε σε δύο νομοθετικές προτάσεις, την ε, Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020 και την Ευρώπη των Πολιτών 2014-2020 πάλι που ήταν το κέντρο από μεγάλο τμήμα της δουλειάς που έκαναν ε, οι προηγούμενες προεδρίες του Συμβουλίου, η Δανία και η Κύπρος. Έχω επίγνωση ότι το Συμβούλιο εξετάζει αυτή τη στιγμή να, το ενδεχόμενο να απαντήσει στις εκθέσεις που υιοθετήσατε πέρυσι ε, στο τέλος του έτους ε, στις προτάσεις της Επιτροπής. Δεδομένου ότι οι συζητήσεις αυτές ε, συνεχίζονται και το Συμβούλιο δεν έχει λάβει ακόμα θέση, δεν μπορώ να συζητήσω πολλά πράγματα μαζί σας σήμερα. Συνολικά ωστόσο έχω επίγνωση ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα που χρειάζεται να συνδιαλλαγούν. Έχω εμπιστοσύνη και προσδοκώ ότι αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με ικανοποιητικό τρόπο τους επόμενους μήνες. Τον περασμένο Νοεμβρίου το Συμβούλιο ε, ε, ε, συμφώνησε εν μέρη στο πρόγραμμα Δημιουργικής Ευρώπης, Creative Europe που περιλάμβανε σημαντικές διατάξεις που έχουν να κάνουν με την ε, διευκόλυνση εγγυήση, που έχουν τον διπλό στόχο της διευκόλυνσης πρόσβασης για το τομέα του πολιτισμού και της δημιουργία, ούτως ώστε να χρηματοδότηση περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και δεύτερον να επιδιώξουν την να επηρεάσουν το, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα για να αξιολογούν τον κίνδυνο στον τομέα της δημιουργία και του πολιτισμού. Αυτή είναι σημαντική η στόχη που αν υλοποιηθούν μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον πολιτισμό και τη δημιουργία. Έχω βεβαίω ταυτόχρονα επίγνωση τη ανάγκη να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση βάσει του πολιετού χρηματοοικονομικού πλαισίου, ούτω ώστε να μπορέσει κάτι τέτοιο να προχωρήσει. Από την έκθεση που εγκρίνατε στην Επιτροπή σα το Δεκέμβριο, βλέπω ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή σα έχουν τι ίδιε ανησυχίε και οι δύο θέλουμε το νέο πρόγραμμα να καλύπτει τι ανάγκε όλων των κλάδων που θεωρούνται πολιτιστικοί και δημιουργικοί και τις ανάγκες όλων των συμμετεχόντων μικρών, μεγάλων, με κερδοσκοπικό ή χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα που δουλεύουν στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργία. Πιστεύω ότι η δουλειά μας στο πρόγραμμα αυτό καθοδηγείται από, τους ίδιους, από τις ίδιες αρχές, που είναι η προώθηση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, η διασφάλιση της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, η εμπλοκή με ένα ευρύ ευρωπαϊκό κοινό και η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις του πολιτισμού και της δημιουργίας, τους, ώστε να μεγαλώσουν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασία και να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ευρωπαϊκό και διεθνέ επίπεδο. Παρά τι διαφορέ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ τη θέσεω του Συμβουλίου και τη θέσεω του Κοινοβουλίου, έχω εμπιστοσύνη στο ότι θα βρεθούν μαζί λύσει. Οι λύσει αυτέ θα εξασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα προσαρμόζεται ε, έγκαιρα στο να μπορούν, ε, θα, θα υιοθετηθεί έγκαιρα, ούτως ώστε να μπορέσουν να υποφεληθούν ο κλάδος και οι δημιουργοί ήδη από το ξεκίνημα του 2014. Η διευκρίνηση της χρηματοδότησης νωρί είναι βασική σημασία και ελπίζουμε ότι αυτό θα λυθεί θετικά στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον άλλο μήνα. Η Προεδρία θεωρεί ότι η Ευρώπη, η Ευρώπη για τους πολίτες είναι μια από τις σημαντικότερες προτάσεις η πρόταση αυτή έχει τη δυνατότητα να φέρει την Ευρώπη κοντά στους πολίτες της και στην παρούσα φάση είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, ο κ. Κένι, ε, δήλωσε πρόσφατα ότι πιστεύει πως η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Παρά τον προπολογισμό 229 εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα 7 χρόνια, το πρόγραμμα αυτό είναι το μόνο που επιδιώκει τη συμμετοχή των πολιτών σε επίπεδο ένωσης και ενισχύει την ανάμνηση. Η Ιρλανδική Προεδρία έχει επίγνωση βέβαια του, των επιπρόσθετων τεχνικού χαρακτήρα θεμάτων χρονοδιαγράμματος που έχουν που, που υπάρχουν, την ανάγκη δηλαδή έγκρισης σε κάποια κράτη-μέλη από τα κοινοβούλια. Καλωσορίζουμε την έκθεση του κ. Τάκουλα, τον οποίο συνάντησα παρεμπιπτόντως σήμερα το πρωί, και που ενέκρινε η Επιτροπή σας τον Νοέμβριο πέρσι. Έχω επίγνωση των δυσκολιών του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την προτινόμενη νομική βάση του θέματος αυτού. Η έκθεση Τάκουλα προτείνει ότι σε ό,τι αφορά την ουσία δεν υπάρχουν ε, μείζονες, ε, σημαντικές, μείζονες διαφορές μεταξύ των στάσεων τη αντιμετώπιση τη πρόταση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Σε πολλέ περιπτώσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο φαίνεται ότι έχουν τι ίδιε ανησυχίε. Ελπίζω και ευελπιστώ ότι οι διαφορέ μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά την νομική βάση δεν θα μας αποτρέψουν από την συμφωνία σε μια πρόταση που έχει σημαντική συμβολική αξία για του πολίτες μας. Οι άλλε προτεραιότητε τη Προεδρία μας είναι να προχωρήσουμε στην πρόταση της Επιτροπής για τι ευρωπαικες πολιτιστικε πολιτιστικέ πρωτεύουσες 2020-2033 και να εξετάσει το θέμα του πολιτισμού ως soft power στις εξωτερικέ μα σχέσεις. Η ιδέα του να γιορτάζουμε τον πολιτισμό σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις είναι πλέον 25 ετών. Έκτοτε πολλά πράγματα άλλαξαν. Ε, μια διυπουργική εκδήλωση έγινε δράση της Ένωσης. Μια ομάδα ε, ειδικών προς επιλογή των πόλεων και, προς την και με στόχο την παρακολούθηση των πολιτιστικών πρωτευουσιών δημιουργήθηκε και σταδιακά ενισχύθη... δημιουργήθηκαν και ενισχύθηκαν κριτήρια. Από την διεύρυνση του 2004 δύο πόλεις από δύο κρατημέλη φιλοξένησαν την εκδήλωση αυτή κάθε χρόνο. Αυτό που δεν άλλαξε είναι αυτό που καθοδηγεί την εκδήλωση αυτή. Το να γιορτάζουμε τον πλούτο και την ποικιλομορφία της κουλτούρας μας και το να φέρνουμε κοντά τους λαούς της Ευρώπης. Το Συμβούλιο καλωσόρισε εν γέννη την τη επιτροπή που στηρίζεται στα θετικά στοιχεία του υφιστάμενου συστήματο ενώ προσπαθεί να διορθώσει τα πλέον αδύναμα. Όπω θα θυμάστε από την ε, έκθεση προόδου που ε, εξέδωσε η Κυπριακή Προεδρία, ο βασικό στόχο ανησυχία ε, που έθεσαν τα κράτη-μέλη σε διάφορα επίπεδα έχουν να κάνουν με ορισμένε διαστάσει των νέων κριτηρίων που εν γέννη ωστόσο έγιναν θετικά δεκτά, την σύνθεση του πάνελ, το να ανοίξουμε το πρόγραμμα σε χώρες που είναι υποψήφιες ή ενδυνάμει υποψήφιες, τον ορισμό των ε, ευρωπαϊκών πολιτιστικών πρωτευουσών και το, τη στιγμή της απονομής ε, του βραβείου Μελίνα Μερκούρη. Ξέρω ότι το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή εξετάζει τα θέματα με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία στις προτινόμενες αλλαγές στην πρόταση. Έχω επίσης επίγνωση ότι ο εισηγητής κ. Σκουρία και οι σκιώδεις εισηγητές εξετάζουν την έκθεσή τους για να την υποβάλουν προς εξέταση στην Επιτροπή. Η Ιρλανδική Προεδρία προσβλέπει στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια έγκαιρη υιοθέτηση της πρότασης αυτής. Η έγκαιρη υιοθέτηση της πρότασης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για την Ιρλανδία, καθότι θα έχουμε το 2020 την πολιτιστική πρωτεύουσα, που θα είναι η πρώτη χρονιά του νέου προγράμματος. Σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό στις διεθνείς σχέσεις και ξέρω ότι αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή σας και την Επίτροπο. Η Ιρλανδική Προεδρία θεωρεί ότι ο πολιτισμός είναι ένα σημαντικό εργαλείο soft power ή soft diplomacy για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των ε, διεθνών, των εξωτερικών σχέσεων και της διπλωματίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο πολιτισμός έχει γνωριστεί ως ε, σημαντικός παράγοντας συνεργασία και με αναπτυσσόμενες και με αναπτυγμένε χώρε. Παρουσιάζοντα την Ένωση ω ε, μια ενότητα με διάφορα πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, ο πολιτισμός μπορεί να βοηθήσει στο να γίνει καλύτερα κατανοητή η Ένωση και οι αξίες τη να, να, και να βελτιωθεί η αμοιβαία κατανόηση με τι χώρε εταίρες. Τα τελευταία χρόνια ε, υπήρξαν, ε, υπήρξε, αυξήθηκαν οι εκκλήσει για την δημιουργία μιας ενός στρατηγικού οράματος του πολιτισμού στην Ευρώπη ειδικά στις εξωτερικές μας σχέσεις. Ξέρω την έκθεση που ετοιμάσατε στην Επιτροπή σας το Μάρτιο του 2011, εξαιρετική έκθεση. Η Προεδρία θέλει να θεωρήσει την, ε, πολιτική πολιτισμού σαν βασικό εργαλείο μας στις εξωτερικές σχέσεις με χώρες όπως η Κίνα. Είχα πάει πρόσφατα στην Κίνα και συνάντησα τον Υπουργό Πολιτισμού της Κίνας που ήταν εξαιρετικά θετικός στην επέκταξη των σχέσεων αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Βασιλείου η Επίτροπος ε, ήταν, είχε επισκεφθεί την Κίνα λίγες εβδομάδες πριν από μένα. Θέλουν πραγματικά οι Κινέζοι να ε, συνεργαστούν στον τομέα αυτό μαζί μας. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ θετική στάση της Κίνας στον τομέα αυτό. Έγιναν ε, πολλές εξετάσεις του θέματος αυτού στο Συμβούλιο και η Επιτροπή περιλαμβάνει την έκθεση για την ε, στρατηγική της Ένωση με την Κίνα στα πολιτισμικά ζητήματα. η Προεδρία θέλει να συζητήσει μια σειρά γενικών αρχών που θα αποτελέσουν τη βάση της ευρωπαϊκής δράσης στον τομέα αυτό. Η Προεδρία καλωσορίζει επίση την πρωτοβουλία τη Επιτροπή να ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση για το Connected για τη TV στο εγγύη μέλλον. Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτε είναι συνδεδεμένοι με smartphone, ταμπλέτε, ε, κομπιούτερ και προσβλέπουν σε ελκυστικό, συνήθως οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Η σύγκληση των παραδοσιακών μορφών ε, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και του ίντερνετ ήδη έχει ξεκινήσει στις ΗΠΑ και σε κάποια κράτη-μέλη της Ένωσης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει η πραγματικότητα το Connected TV. Η Προεδρία θεωρεί ότι, είναι, αυτό, ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό με πάρα πολύ μεγάλες πολιτισμικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής σας, ιδιαίτερα την πρωτοβουλία της κυρίας Καμέρε Βέρτ για τι τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με το Connected TV. Ξέρω ότι ο, συνάδελφο, ο συνάδελφος θα εξετάσει το θέμα αυτό για να δούμε κατά πόσο μπορεί να συνεργαστούμε το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στον τομέα αυτό. Κλείνοντα, σα ευχαριστώ κύριε Πάκ για την ευκαιρία που μου δώσετε να παρουσιάσω τι βασικέ μα προτεραιότητε. Προσβλέπουμε στη συνεργασία εξ του Συμβουλίου με την Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευση και Παιδεία και την Κομισιόν του επόμενου μήνε κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα, με στόχο να πετύχουμε έγκαιρη έγκριση των σημαντικών νομοθετικών κειμένων που έχουμε μπροστά μα. σας. Να σα προτείνω επίσης να εξετάσετε και το πρόγραμμά μας δραστηριοτήτων στις Βρυξέλλες με εξαιρετικά καλές παραστάσεις από την αφρόκρεμα της Ιρλανδικής κουλτούρας στους επόμενους μήνες. Να τονίσω επίσης ότι ότι οι δραστηριότητες αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει από τον ε, περασμένο Μάιο και νομίζω ότι ορισμένοι από εσάς τους έχετε ήδη δει. Ευχαριστώ πολύ για την ε, προσοχή σας. Ευχαριστώ εγώ κύριε Υπουργέ. Πριν ε, δούμε το πρόγραμμα, θα μπορούσαμε κάλλιστα να δούμε εδώ μέσα στο κοινοβούλιο τι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες ε, εικόνες, φωτογραφίες που είναι ε, Ιρλανδικές φαίνεται και κοσμούν τους τοίχους του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις, έχουν όντως ξεκινήσει πάρα πολλά πράγματα να γίνονται. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε ούτω ή άλλω πολλά Ιρλανδικά δρόμενα και βεβαίω και στην πόλη θα υπάρχουν πολλέ δραστηριότητε. Λοιπόν, πριν ε, ξεκινήσουμε την ε, συζήτηση, να δώσουμε τον ε, λόγο στον Υπουργό Ring, αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού. Thank you very much, Chairperson. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Είναι χαρά μου που είμαι σήμερα εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευση για να παρουσιάσω τι προτεραιότητε για τον αθλητισμό τη Ιρλανδική Προεδρία για το επόμενο εξάμεινο. Όπω ξέρετε, η Ιρλανδία είναι η πρώτη χώρα της, ε, του, της Προεδρίας των, ε, του Τρίο που ε, αποτελείται από τη Λιθουανία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα που έχει ένα πρόγραμμα που ξεπερνά όλα τα Υπουργεία και θέλει να προωθήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας η Ιρλανδία θεωρείται ε, κράτος αθλητών και ελπίζουμε ότι αυτή η παράδοση μαζί με την εμπειρία που έχουμε θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια επιτυχή προεδρία για τον τομέα του αθλητισμού. Είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή μαζί σας τον τελευταίο χρόνο με κάποιους από εσά για να συζητήσουμε θέματα αθλητισμού και βεβαίω περιμένω να κάνω μια ζωντανή συζήτηση και σήμερα. Γιατί όντω η συμβολή του Κοινοβουλίου είναι σημαντική για τον τομέα αυτό μια που υπάρχει και η ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. Υπάρχει ε, υπάρχουν πολλά οικονομικά, κοινωνικά ωφέλη από τον, από τον αθλητισμό και βεβαίω είναι σημαντικό να συνοδοποιήσουμε την σημασία του αθλητισμού για την κοινωνική ανάπτυξη και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο αθλητισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της υγείας και της ευημερία των πολιτών μας και δίνει και την αίσθηση του ότι ανήκουν, ε, σε κάποιο, ανήκουν κάπου όλοι αυτοί που ακολουθούν ε, τέτοιες δραστηριότητε και ε, εξασκούνται. Προσπαθούμε λοιπόν να ενισχύσουμε την συμμετοχή των πολιτών στις, σε αθλητικές δραστηριότητες η ε, επιτυχία των δικών μας αθλητών ε, έχει να κάνει και με τον δίκαιο ε, ανταγωνισμό και βεβαίως μπορεί να ενισχύσει και την συμμετοχή άλλων. Οι αθλητές μας είναι υποδείγματα για τους νέους μας και αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη να προστατεύσουμε την ακαιρεότητα του αθλητισμού. Κανένα δεν μπαίνει στον αθλητισμό έχοντα ω πρόθεση να εξαπατήσει. Ξέρουμε βεβαίω ότι αυτό συμβαίνει. Ε, και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι θεμελιώδει ιδέε και οι αξίε του αθλητισμού θα προστατεύονται και δεν θα χαθούν στην, ε, στο δρόμο, στην προσπάθεια. Ε, βεβαίω, ο αθλητισμό συμβάλλει σημαντικά και στην ευρωπαϊκή οικονομία και όντω ενισχύει και την ανάπτυξη και την απασχόληση. Εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την ευημερία. Και αυτό βοηθά και στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής 2020. Ε, Γιατί, ενώ μάλλον ε, ε, εννοούμε ότι είναι σημαντικό το θέμα του αθλητισμού για τα κράτη-μέλη, η νέα ευρωπαϊκή πολιτική επιτρέπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη να συνεργαστούν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντο και να μοιραστούν τι βέλτιστε πρακτικέ. Επίση, μα δίνει τη δυνατότητα να μιλούμε με μία φωνή σε διεθνέ επίπεδο ιδιαίτερα σε τομεί όπω η αντιμετώπιση ε, του ντόπινγκ, που είναι πραγματικά ιδιαίτερο ανησυχητικό φαινόμενο, καθώ επίση και η αντιμετώπιση τη διαφθοράς στον αθλητισμό. Από κοινού λοιπόν μπορούμε να προσπαθήσουμε ώστε να βελτιώσουμε και να προστατεύσουμε την ακαιρεότητα του αθλητισμού, να αποτρέψουμε την ξαπάτηση σε όλα τα επίπεδα και να ενισχύσουμε, να προωθήσουμε τον υγιή αθλητισμό. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε πολλέ προτεραιότητε κατά τη διάρκεια τη προεδρία μα. Η Προεδρία μα θέλει να εξασφαλίσει την εφαρμογή του πρώτου ε, ε, ε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον αθλητισμό αποκοινούμε την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη και με την στήριξη βεβαίω των ε, εταίρων μα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι, οι ε, προτεραιότητέ μα έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση του αθλητισμού, με θέματα προστασία τη εκαιρεότητα του κλάδου το Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει την σημασία των, των, της καριέρας που μπορεί να κάνει ένας αθλητής και αυτό θα αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες των, της Προεδρίας μας. Πολλές φορές οι αθλητές έχουν να, έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις ε, στο συνδυασμό της αθλητικής τους ε, πορείας με την ε, εργασία τους. Για να επιτύχουμε λοιπόν το, το ανώτερο επίπεδο αθλητισμού πρέπει προφανώς να ε, υπόκειται κανείς σε τεράστιο ανταγωνισμό και αυτό ε, πρέπει να το δούμε και στα πλαίσια των εργασιακών ε, δραστηριοτήτων που έχει ο καθένα. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε την περίπτωση όπου αθλητές αναγκάζονται να διαλέξουν ανάμεσα στον, στην εργασία τους ή στον αθλητισμό. Με βάση και τα διαφορετικά συστήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε όντω να έχει προσθέμενη αξία στην προσπάθειά τη να αντιμετωπίσει το θέμα τη ε, καριέρα, τη επαγγελματική ε, δραστηριότητα των αθλητών. Και αυτό έχει να κάνει και με πολλά από τα σημεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Ευρώπη 2020. Γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε τους, ε, αθλητές, ε, τους πρώτα στον αθλητισμό. Το Νοέμβριο του 2012, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον αθλητισμό και την εκπαίδευση σε μια, α, α, κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για τον αθλητισμό έτσι ώστε να ενισχυθεί η υποστήριξη των αθλητών ώστε να μπορούν να διατηρήσουν και τι επαγγελματικέ του δραστηριότητε. Η Ιρλανδική Προεδρία λοιπόν θα προετοιμάσει ένα, ε, μια δέσμη ε, συμπερασμάτων του Συμβουλίου έτσι ώστε να μπορούν να ε, περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία αυτά και του πολυαθλητισμού και της επαγγελματική καριέρας και της εκπαίδευσης. Το θέμα της οικονομικής συνεισφορά ε, αλλά και τη χρηματοδότηση του αθλητισμού είναι από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Προεδρία και αποτέλεσε προτεραιότητα και, της προεδρίας, και του τρίου των Προεδριών. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλά στοιχεία μέσω διαφόρων μελετών που έγιναν πρόσφατα και ο, 173 ε, δισεκατομμύρια είναι η συνεισφορά του αθλητισμού στην, στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μιλούμε δηλαδή για 2,12% ε, και 2,12% απασχολούμενο στον αθλητισμό ε, στην Ευρώπη πάντα. Η οικονομική κρίση βεβαίω έχει τεράστιε επιδράσει στην, ε, στην χρηματοδότηση πολλών δραστηριοτήτων, μεταξύ αυτών και ο αθλητισμό. Πρέπει βεβαίω να ενισχύσουμε τη βιώσιμη χρηματοδότηση του αθλητισμού 7 και 8 Μαΐου θα γίνει μια συνάντηση στην, ε, των υπευθύνων ε, περιαθλητισμού στην, στο Δουβλίνο για να συζητήσουν τα θέματα αυτά. Η ομάδα αυτή εμπειρογνωμόνων ε, συνέστησε ότι πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί διαφύλαξης της χρηματοδότησης του αθλητισμού έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τις υπόλοιπες προεδρίες, ώστε να, να μελετήσουν το θέμα αυτό ακόμη πιο προσεκτικά. Οι, οι οικονομικές συνέπειες ε, στον ε, αθλητισμό, το πώς χρηματοδοτείται ο αθλητισμός, και κάποιε από τι οικονομικέ προκλήσει που έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδο είναι θέματα πολύ σημαντικά. Θέλουμε λοιπόν να ε, ανταλλάξουμε τι βέλτιστε πρακτικέ για το πώ τα κράτη-μέλη και οι διεθνεί οργανισμοί χρηματοδοτούν τον αθλητισμό και πώ έχουν ε, συνεργαστεί ώστε να δημιουργήσουν έναν ε, μηχανισμό χρηματοπιστωτική οικονομική αλληλεγγύη για τον αθλητισμό. Βεβαίω εμπλέκονται σε όλο αυτό και οι διάφορε αθλητικέ ενώσει και σύλλογοι η αντιμετώπιση και τη ανεργία είναι κάτι για το οποίο η Ιρλανδική Προεδρία ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Οι μεγάλες προκλήσει που έχει να αντιμετωπίσει ο αθλητισμός είναι η καταράκωση της, της ε, του λόγω διαφόρων ε, συμβάντων που έχουμε παρατηρήσει και που είναι ε, ανάντια σε όλε τι αξίε του ε, αθλητισμού. Όλα αυτά λοιπόν η Ιρλανδική Προεδρία θα τα προωθήσει. Θα παρακολουθούμε στενά όλε τι διεθνεί εξελίξει ό,τι αφορά το στήσιμο των παιχνιδιών. Στο Συμβούλιο η Ιρλανδική Προεδρία θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει μια απόφαση του Συμβουλίου ε, με, μια δημοκρατική εντολή για την Κομισιόν, ώστε να υπάρξει ένα συμβούλιο ε, που θα ασχολείται ακριβώ με το θέμα των, του στησίματο των παιχνιδιών. Πρέπει λοιπόν όλοι οι εταίροι να συνεργαστούν ώστε να, ε, προσπαθ... να καταφέρουμε να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο όλων αυτών στον αθλητισμό. Ω Προεδρία θέλουμε να προετοιμαστούμε για την πέμπτη διεθνή διάσκεψη των Υπουργών και των Ανώτερων Αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για την γυμναστική και τον αθλητισμό που θα γίνει στο Βερολίνο ε, τον ε, Μάιο διατηρώντα πάντα την ακαιρεότητα του αθλητισμού. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τον αθλητισμό ε, απέναντι στο ντόπινγκ, που είναι τελείω αντίθετο ε, με τι αρχέ του αθλητισμού, του δίκαιου ανταγωνισμού, ε, τη ειλικρίνεια. Ο αθλητισμό προάγει τον θεμητό ανταγωνισμό και ε, τα κρούσματα ντόπινγκ μπορεί όντω να αποτρέψουν του νέου να συμμετέχουν σε αθλητικέ δραστηριότητε. Το ντόπινγκ επίση αποτελεί τεράστια απειλή και για την ε, δημόσια υγεία και μπορεί να έχει και μακροπρόθεσμε ε, παρενέργειε στην υγεία των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει τιμωρία και βεβαίω πρέπει να υπάρχει και καλύτερη εκπαίδευση των αθλητών για να, μην, να, να του αποτρέψουμε από το να παίρνουν τέτοιε απαγορευμένε ουσίε. Από το 1999 προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ντόπινγκ στον αθλητισμό. Ε, το, ο κώδικας ε, για το anti-doping ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο γιατί θέτει ακριβώς τους κανόνες για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτό. Είναι λοιπόν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μία φωνή στον τομέα του anti-doping. Μόνο όταν συνεργαστούμε μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό και με συνεκτικό τρόπο θα πρέπει αυτό να γίνει και στα πλαίσια της WADA. Ε, ή τα κρατημέλη πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και στη Γουάντα από το 2013 και μετά, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερη συνέχεια στην εκπροσώπηση τη ευρωπαϊκή θέση. Η Ιρλανδία θα εκπροσωπήσει το, το τρίο των Προεδριών για του επόμενου 18 μήνε και βεβαίω προσβλέπουμε στο να προσφέρουμε τη δική μα εμπειρία στον τομέα αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και εμεί την αντιμετώπιση του ντόπινγκ στην, στον αθλητισμό. Θα υπάρξει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή θέση για την Γουάντα. Η ευρωπαϊκή ε, θέση θα παρουσιαστεί από την Προεδρία στο, στη συνεδρίαση της Γουάντα 12 και 13 Μαΐου και η Ιρλανδική Προεδρία θα προετοιμάσει μια συντονισμένη ε, παρέμβαση ευρωπαϊκή για, την, ε, για τον κώδικα για το αντιντόπινγκ με συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα. Εξεκολουθούν να υπάρχουν λοιπόν θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αφορά τον ντόπινγκ και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να, βρούμε κάποια λύση για όλα αυτά τα προβλήματα έτσι που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από όλου. Βασικό στόχο τη Ισλανδική Προεδρία θα είναι να καταλήξουμε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάνω στι προτάσει τη Κομισιόν για ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον αθλητισμό. Βεβαίω ο αρμόδιο υπουργό θα είναι ο Υπουργό ε, Εκπαίδευση ε, και το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί. Πολλά κράτη-μέλη υποστήριξαν την ε, δημιουργία ε, μιας Ευρωπαϊκής ημέρας για τον ε, αθλητισμό που θα μπορέσει να προωθήσει διάφορες ε, φυσικές δραστηριότητε. Και βεβαίω αυτή η πρόταση είναι αρκετά καλή, αρκετά ενδιαφέρουσα, έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε όσου δεν κάνουν διάφορε δραστηριότητε αθλητικέ στη ζωή του να το πράξουν και να τι ενσωματώσουν στο καθημερινό του πρόγραμμα. Είναι εύκολο να εμπλακεί κανεί στον αθλητισμό και αφορά όλου ανεξαρτήτω ηλικία. Το 2013 ξέρετε ότι είναι το ευρωπαϊκό έτος του πολίτη. Έχει... Ο αθλητισμό μπορεί λοιπόν να παίξει ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά και την κοινωνική συνοχή και κυρίω μεταξύ των νέων. Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα ο αθλητισμό θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα μέτρα για την πρόθεσή του. Σα ευχαριστώ και ευχαρίστω να απαντήσω στι ερωτήσει. Εγώ ευχαριστώ. Μπορούμε τώρα να συζητήσουμε και τις ε, δύο αυτές παρουσιάσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Υπουργούς ε, για, την, ε, για τις ομιλίες τους. Πολύ περιεκτικές και σαφέστατες. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω προς τον κύριο Ρίνγκ. Το πρώτο ερώτημα αφορά τα στημένα παιχνίδια θα γνωρίζετε το γεγονός ότι εμείς έχουμε ήδη ε, ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Έχουμε δεσμευτεί ε, πολύ περισσότερο τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι σαφές για όλους μας ε, πλέον ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ σοβαρό και δύσκολο πρόβλημα. Κάναμε και μία ακρόαση για αυτό το θέμα πριν από τα Χριστούγεννα. Κάποιοι εμπειρογνώμονες μας είπαν πόσα πολλά πράγματα διακυβεύονται. Το ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω, μια και μιλάτε με τόσο ζήλο για την ε, καταπολέμηση του ντόπινγκ, θα τοποθείτε με τον ίδιο τρόπο κατά της διαφθοράς ε, και του στισίματος των παιχνιδιών ε, στον αθλητισμό, γιατί είναι εξίσου σοβαρά προβλήματα και πώς μπορεί το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο να εργαστούν επιπρακτικών λύσεων. Ξέρω ότι έχουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Σύμβαση κατά του ντόπινγκ, αλλά ε, στην πράξη τι πρέπει να γίνει και ποια είναι τα σχέδιά σας ως προς αυτό. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους υπουργού για τις παρεμβάσεις τους. Ακούσαμε με ιδιαίτερη χαρά, κύριε Υπουργέ, κύριε Τένιχαν, ότι ε, θέλετε να προωθήσετε το πρόγραμμα για τους, για τους πολίτες, Ευρώπη για τους πολίτες και εμείς ε, το προωθήσαμε αυτό, ανεξάρτητα βεβαίως από τις ανησυχίες και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την νομική βάση. Εμείς βεβαίως ε, χαιρόμαστε που θέλετε να προωθήσετε και τις δικές μας προτάσεις. Χαίρομαι ότι στο, γιατί στο τέλος θα καταφέρουμε, ελπίζω, να καταλήξουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα Οπότε τελικά το πρόβλημα της νομικής βάσης νομίζω ότι δεν θα είναι το ουσιώδες. Χαίρομαι που θέλετε κι εσείς να προωθήσετε δυναμικά την Ευρώπη για τους πολίτες. Ε, για τον αθλητισμό να πω κάτι κύριε Ρίνγκ. Ε, ξέρετε ότι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο ασχοληθήκαμε πολύ ε, και με την διπλή εκπαίδευση, κατάρτιση Αναφέρατε κι εσείς ε, κάποιες ε, εκθέσεις που υπάρχουν και πρέπει όντως να φροντίσουμε έτσι ώστε οι επαγγελματίες αθλητές να μην είναι μόνο καλοί στον, στον τομέα τους αλλά να έχουν ε, μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση και βεβαίως επαγγελματική κατάρτιση. Αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά το, το πρόβλημα να έχουμε πολύ καλές ιδέες αλλά στην πράξη τελικά να μην γίνεται κάτι. Οπότε είναι αξιέπαινο πραγματικά το ότι εσείς θέλετε να δραστηριοποιηθείτε για τον τομέα αυτό. Ξέρουμε βεβαίως ότι η, ε, το να υπάρξουν, ε, όταν υπάρχουν νομικές, νομικά δεσμευτικές ε, διατάξεις για τα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη αντιδρούν. Θα μπορούσατε να φανταστείτε, ας πούμε, να σκεφτείτε ότι στο, στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν ίσως να αυτοϋποχρεωθούν να κάνουν κάτι ακριβώς ό,τι αφορά την διπλή εκπαίδευση, κατάρτιση των αθλητών. Να κάνουν πολύ περισσότερα δηλαδή από μόνα του. Υπάρχουν πολλά κρατημέλη που έχουν πολύ καλά παραδείγματα να δείξουν, ευέλτιστε πρακτικέ, συγκεκριμένα μοντέλα, τα οποία θα μπορούσαν να τα μιμηθούν και άλλα κρατημέλη. Αν λοιπόν υποχρεωθεί το κάθε κράτο μέλο από μόνο του να, να δράσει περισσότερο στον τομέα αυτό, σε εθνικό επίπεδο, ε, είτε α πούμε με των κειμένων, και εμεί βεβαίω ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε λιγότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς αυτό, νομίζω ότι θα ήταν ένα βήμα προς τα εμπρός. Δεν ξέρω, θα μπορούσατε να φανταστείτε να κινηθούμε προς μια τέτοια κατεύθυνση, μια δηλαδή υποχρέωση των κρατών μελών, χωρίς όμως αυτή η υποχρέωση να είναι ευρωπαϊκή, να είναι μια υποχρέωση που θα επιβάλλουν τα κράτη-μέλη από μόνα τους στον εαυτό τους. Ο κύριος ευχαριστώ πρόεδρε και να ευχαριστήσω εγώ τους Ιρλανδούς υπουργού που ήρθαν εδώ για να μας παρουσιάσουν με εξαντλητικό τρόπο τις προτεραιότητες τους. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τους προλαλήσαντες ό,τι αφορά τον αθλητισμό των νέων. Δηλαδή, είναι, είναι χρήσιμη η αθλητική δραστηριότητα, αλλά τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν. Κάτι που συχνά δεν συμβαίνει. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πιο διεξοδικά, λόγοντα και του, των μικρών δυνατοτήτων που έχουμε νομοθετικά, πώς μπορεί να, να δείτε αυτό το πράγμα. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι αναφορέ που κάνετε για το ντοπάρισμα και τα στημένα παιχνίδια που πραγματικά καταστρέφουν την ε, αθλητική, τον αθλητικό πολιτισμό, την κουλτούρα του αθλητισμού και πρέπει να καταπολεμηθούν πιο, πιο συγκεκριμένος τόσο τι μπορεί να γίνει διότι δυστυχώς ε, σε ό,τι αφορά ιδίω τα στημένα παιχνίδια ξέρουμε ότι το θέμα αυτό είναι κάτι που ξεπερνά τα όρια όχι μόνο των κρατών μελών αλλά και της Ευρώπης μερικές φορές. Δύο παρατηρήσεις. Άκουσα πρώτα να γίνεται λόγος και χάρηκα γι' αυτό για τη διασφάλιση της γλωσσικής και πολιτιστικής διαφορετικότητας. Είσαστε και υπουργό ε, τη Ιρλανδικής γλώσσα. Το πρωί σήμερα μιλούσαμε για μια πρωτοβουλία που ξεκινά στην Επιτροπή Πολιτισμού για τις γλωσσικέ μειονότητες. Και από την άποψη αυτή ωστόσο δεν έχουμε πολλές εξουσίες. Δεδομένου ωστόσο ότι σα ενδιαφέρει ιδιαίτερα, θα ήθελα να ακούσω λίγο περισσότερα πράγματα από εσά για αυτό το σημαντικότατο ζήτημα. Κάθε γλώσσα είναι ένας πολιτισμός το να χάσουμε μία γλώσσα, χάνουμε και ένα κομμάτι του πολιτισμού της Ευρώπης, κάτι βασικό. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τους νέους είναι ότι, όλο, ότι διαβάζουν όλο και λιγότερο οι νέοι. Έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε κάπως την, την ανάγνωση των βιβλίων από τους νέους, ίσως και με νέες τεχνολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ε, ευχαριστώ πολύ που δώσατε και το βήμα ε, στους συναδέλφους ε, από την Ιρλανδία και φίλους μου εδώ και πολύ καιρό. Έχετε μιλήσει πολλές φορές για τις προσδοκίες σας από την Ιρλανδική Προεδρία. Είστε εδώ τώρα. Είμαι βέβαιος ότι οι Υπουργοί θα κάνουν ό,τι μπορούν για να προωθήσουν πολλά ζητήματα τα οποία, για τα οποία μας μίλησαν την τελευταία μισή ώρα. Και επίση ε, μπορώ να πω ότι όχι, ελπίζω ότι όχι μόνο τα λόγια τους αλλά και οι πράξεις τους ε, ήταν ε, πραγματικά πολύ ένθερμες και υπέρ του αθλητισμού. Το είδαμε αυτό και στις ομιλίες σας σήμερα. Ο Υπουργός Ντένιεν αναφέρθηκε στο θέμα του προγράμματος του πολιτισμού. Θέλουμε όλο και περισσότερη χρηματοδότηση τη μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα αυτό. Μιλάμε για την απασχόληση, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ότι είναι μια ευκαιρία για μας να δημιουργήσουμε θέσει απασχόλησης ε, και να δούμε τι πλεονεκτήματα έχουμε στο ίδιο το πρόγραμμα για τον πολιτισμό. και το λέω αυτό σε σχέση με το πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο, πόσο περισσότερα μπορούμε να επιτύχουμε για το πρόγραμμα του πολιτισμού και ελπίζουμε να μην θυσιαστούν ε, στην ε, ολόκληρη, στη μάχη που πρέπει να δώσουμε για τη χρηματοδότηση άλλων τομέων. Ελπίζουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί όπως το αξίζει. Ε, προς τον κύριο Ρίγκ, ο οποίος κάλυψε πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν πολύ και τα έχουμε συζητήσει εδώ πολλές φορές. Ε, ε, τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε και ένα πρόγραμμα για τον αθλητισμό που θα χρηματοδοτηθεί για πρώτη φορά κατά το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι ένας από τους τομείς για τους οποίους και εγώ και άλλοι έχουμε πολλές φορές πει πόσο μεγάλη είναι η σημασία των τοπικών παραγόντων ε, ακόμη και στο χαμηλότερο επίπεδο, στη χαμηλότερη βαθμίδα και πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε μέσω μέτρων που θα, που θα λάβουμε για να υπάρξει καλύτερη χρηματοδότηση ε, του αθλητισμού σε αυτό το επίπεδο, στο τοπικό επίπεδο, στο επίπεδο της χαμηλότερης βαθμίδας. Είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε, το συζητάμε εδώ και δύο χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ και μπορείτε να βασιστείτε στη συνεργασία μας για τους επόμενους έξι μήνες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κώστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους Υπουργούς για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων του προγράμματος. Εύχομαι να είχαμε ήδη την ευκαιρία να συναντηθούμε τον Υπουργό Πολιτισμού και να δούμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στο Ιρλανδικό πρόγραμμα ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα, καθώς και ο αθλητισμός. Νομίζω ότι αυτό δίνει περαιτέρω ανάπτυξη στην Ευρώπη που λαμβάνει όλους υπόψη της. Ως εισηγήτρια για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη εύχομαι να υπάρξει καλή συνεργασία με το Συμβούλιο και δυνατότητα να υπάρξει εξαιρετική συμφωνία που θα λαμβάνει και υπόψη την σύνθετη, την αναζήτηση μάλλον αυτού, αυτής της σύνθετης συμφωνίας στο εσωτερικό της Επιτροπής και με το Συμβούλιο για το ζήτημα αυτό. Η έκθεση που ανέφερε και ο Υπουργό είναι καρπός μια ευρεία ε, συνένεσης. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη. Να σας πω ωστόσο ότι από την άλλη πλευρά σε ό,τι με αφορά όταν είχα κάνει την έκθεση είχα λάβει υπόψη πολλέ από τις διαστάσεις που είχαν περάσει από αυτή την μερική συμφωνία του Συμβουλίου των Υπουργών το, Μάρτιο το Μάιο Πέρσι, συγγνώμη, Κάποιε από τις ανησυχίε που είχαν εκφραστεί εκεί περιλαμβάνονται στην έκθεση. Ελπίζω αυτό να το καταλάβετε. Να υπογραμμίσω τρία πράγματα που θα τα δούμε και θεσμικά κατόπιν. Πρώτον, τη βούληση να προχωρήσουμε προς ένα πρόγραμμα πλαίσιο με διακρίνοντας ωστόσο αυτό που είναι πολιτισμός, κληρονομιά και ενόψη και διάκριση των μη κυβερνητικών, των μη κερδοσκοπικών, της μη κερδοσκοπικής διάστασης σε σχέση με τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Διατηρώντας ε, ταυτόχρονα το θέμα της governance ε, που για το Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό. Στον τομέα αυτό πιστεύουμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο ρόλο για την παρακολούθηση και τούτο να γίνει και με κατεξουσιοδότηση πράξη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διατήρηση της χρηματοδότησης της, για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη σε σχέση με την κατάσταση της τρέχουσας ε, επταετίας ε, ενώ παραμένουμε κάτω από το 1% στον προπολογισμό του, του πολιτισμού έχουμε πολύ ε, μεγαλύτερα προγράμματα. Αυτό έχει πολιτικές επιπτώσεις. Θα ήθελα επίσης να ακούσω την άποψή σας και να βρούμε και μια συμφωνία και για τον τρόπο με τον οποίο με τους συναδέλφους βρήκαμε μια πρόταση για το νέο χρηματοοικονομικό εργαλείο που περιλαμβάνει το Ingrance με μιλήσατε για την δυνατότητα χρησιμοποίησης ε, ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Το εύχομαι, αλλά εμεί έχουμε θέσει και άλλες προϋποθέσεις που μπορούν να μετατρέψουν το εργαλείο αυτό προς πελάσιμο και να του επιτρέψουν να δημιουργήσει καλύτερα μια σειρά, ένα πλαίσιο ε, χρηματοδότησης ε, του πολιτισμού. Ελπίζω στο σημείο αυτό να βρούμε μια συμφωνία, όχι καθυστερημένα. Ευχαριστώ Σίλβια. Ο κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμη Υπουργέ. Υποθέτω ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά την ε, σημασία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ε, της Διαβίου Μάθησης. Ειδικά για τους νέους, ε, ας πούμε το Grundvik, το Erasmus, όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Μέσω λοιπόν αυτής της πολύ ενεργής, ενεργούς ε, πρωτοβουλίας, νομίζω Κύριε Μπεκέρ, συγγνώμη, αλλά δεν μιλούμε για τα προγράμματα, μιλούμε για την ε, ευρωπαϊκή ε, ηθαγένεια και τον αθλητισμό. Την ερώτησή σας μάλλον πρέπει να την ε, θέσετε στο επόμενο πάνελ. Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ. Ο κύριος Κουρία. Ευχαριστώ. Πατώτε. Σύντομα. Ευχαριστώ τους υπουργούς για την παρουσία τους μας παρουσίασαν το πρόγραμμά τους. Θα ήθελα, όπως και κάποιος άλλος συνάδελφος ανέφερε, να καταλάβω αν ανάλογα με την αρμοδιότητα που έχουν, είναι διαθέσιμοι να δουλέψουν για την αύξηση του προϋπολογισμού... των πόρων δηλαδή, που θέτει η Ένωση στα θέματα που συζητούμε σήμερα το απόγευμα. και σε περίπτωση δυσκολία ε, εξέβρεση πόρων, ποια άλλα εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουμε για πρώτη φορά σε κοινοτικό επίπεδο να φανταστούμε την δημιουργία πόρων που θα μπορέσουν να καλύψουν τα προγράμματα που μιλούμε και με παρέμβαση ιδιωτών. Με ένα είδος ε, χορηγίας ποντινά. Εμείς έχουμε ακούσει πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες. Εμείς δουλεύουμε και στο επίπεδο της πολιτιστικής ε, αθλητικής ε, προσφοράς. Αν μείνουμε όμως ε, κολλημένοι στα οικονομικά δεν θα κατορθώσουμε να φέρουμε το σκάφος σε ασφαλή λιμένα. Θα ήθελα λοιπόν να δω κατά πόσον η Ιρλανδική Προεδρία θα είναι σύμμαχός μας στο Συμβούλιο για να βελτιώσει την οικονομική διάσταση της χρηματοδότησης του πολιτισμού που μειώνεται από τη βλέπουμε. Ενώ εμείς είχαμε εικόνα ότι θα, θα αυξάναμε λίγο τον προπολογισμό. Η Ιρλανδική Προεδρία θα στοιχηματίσει στον αθλητισμό και στον πολιτισμό ως πραγματικό πόρο της Ένωσης. Ευχαριστώ. Οπότε τώρα έχουν οι υπουργοί την άνεση να απαντήσουν. Ποιο θέλει να ξεκινήσει. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλές οι ερωτήσεις, ε, κύριε Λάκη και κύριο Φοντάνα. Πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα. Όντως, ε, έχω ιδιαίτερο ζήλο για το να κλέβει κανείς ε, το ντόπινγκ στον αθλητισμό, γιατί στον αθλητισμό πρέπει να είναι ίσοι όταν ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Και σε σχέση τώρα με το ντόπινγκ το νέο βιολογικό διαβατήριο που μπορεί να γίνει στον αθλητισμό είναι ένας πολύ καλός τρόπος προσέλκυσης ε, ανθρώπων στον αθλητισμό και ένας, και τρόπος να διακοπεί το ντόπινγκ. Πρέπει όμως, επειδή θα είναι κάτι δύσκολο, να συνεργαστούμε. Γιατί και το στήσιμο των παιχνιδιών είναι κάτι το οποίο ζημιώνει ε, τον αθλητισμό. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει ε, όλες όλοι οι δομές πρέπει, όλες οι δομές πρέπει να συνεργαστούν ε, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερους θεατές και τους νέους, γιατί όταν οι νέοι ε, κλέβουν και ντοπάρονται, αυτό είναι πάρα πολύ επιβλαβές για τον αθλητισμό. Επαναλαμβάνω, πρέπει όλοι να συνεργαστούμε. Αυτή είναι η δική μου δουλειά στους επόμενους έξι μήνες να προσπαθήσουμε όλοι να συμπορευτούμε σε αυτή την προσπάθειά μας. Κυρία ε, Καμερβέρτ, θέσατε ένα θέμα για τους νέους και την εκπαίδευση. Γίνεται ιδιαίτερη δουλειά στον τομέα αυτό από την ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων. Ε, συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα στην Ιρλανδία. Ελπίζω και εγώ να πάω να τους μιλήσω. Νομίζω ότι η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, την οποία θα ενθαρρύνει και η ομάδα. Θα έχω τη δυνατότητα δυνατότητα να τους μιλήσω την επόμενη εβδομάδα και ελπίζω να υπάρξουν και συμπεράσματα του Συμβουλίου μέχρι το τέλος της Προεδρίας μας ε, ως προς αυτό. Κύριε Κέλλη, με ρωτήσατε για την ε, ε, σωστή χρηματοδότηση, μιλήσατε για το ντόπινγκ, μιλήσατε ε, για το στήσιμο και μιλήσατε και για, τους, για τον, τοπικό και χαμηλής βαθμίδας αθλητισμός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο να το υποστηρίξουμε, γιατί μερικές φορές ξεχνάμε στον αθλητισμό και θεωρούμε ότι υπάρχει μόνο η αφρόκρεμα στον αθλητισμό, χωρίς όμως τους εθελοντές, τους δεν θα είχαμε τέτοιου είδους αφρόκρεμα στον αθλητισμό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να τους προστατεύσουμε και να εξασφαλίσουμε σχετική χρηματοδότηση. Χαίρομαι πολύ και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη σε σχέση με την εβδομάδα του αθλητισμού. Είναι και αυτό σημαντικό. Είναι σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση, δηλαδή ότι όλο ο κόσμο πρέπει να μπορεί να συμμετέχει και να είναι επίση διασκέδαση, να μην είναι μόνο... Ε, ε, ανταγωνισμός να ε, μπορεί να είναι απλώς ε, διασκέδαση. Όσο περισσότερο περικόπτουμε τη χρηματοδότηση του αθλητισμού, τόσο λιγότερα νοσοκομεία έχουμε, τόσο λιγότερους γιατρούς, τόσο λιγότερες νοσοκόμες και πρέπει να πείσουμε ότι τα χρήματα για τον αθλητισμό, όταν δαπανώνται στον αθλητισμό, δαπανώνται καλώς. Ο κύριος Κούρια, μιλήσατε για την ιδιωτική χρηματοδότηση. Σε σχέση με τη χρηματοδότηση της δαπάνης για τον αθλητισμό, είναι ό,τι χρήματα μπορούμε να δώσουμε στον αθλητισμό, πρέπει να τα δώσουμε. Και αν ο κόσμος θέλει ιδιωτικά να συνεισφέρει, τόσο το καλύτερο. Πρέπει να έχουμε προτεραιότητε. Ε, πρέπει ο κόσμος να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τον αθλητισμό και το λέω αυτό και σε χαμηλότερο επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τον κόσμο σε νεαρή ηλικία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντένιαν. Ε, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πακ. ευχαριστώ και τον ε, συνάδελφό μου για τις ε, πολύ καλές απαντήσεις του. Κυρία Καμερβέρ, μπορώ να σας πω Γνωρίζετε ότι η αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου ασχολείται με το θέμα αυτό. 26 Νοεμβρίου ε, τοποθετήθηκε επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεχίζονται λοιπόν οι συζητήσεις. Πρόκειται να καταλήξει σε μία θέση το Συμβούλιο. Δεν μπορώ βέβαια να το συζητήσω αυτή τη στιγμή με το Κοινοβούλιο, αλλά από έχω ακούσει και βάσει της ενημέρωσής μου δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι θα μπορέσουμε, όπως είπε και η κυρία Πακ, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα είναι υποφελής για όλους και μενα βεβαίως ε, ε, είναι πολύ σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και γι' αυτό, και γι αυτό μάλιστα ε, γι' αυτό ακριβώ μιλούσε και η συνθήκη της Λισαβόνα, το να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τις, ε, για τις προεκλογικές μας εκστρατείες ευρωεκλογές. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που ένα τόσο καλός άνθρωπος ήταν το αποτέλεσμα αυτής της προεκλογικής εκστρατεία. Αλλά αυτή ήταν η εκστρατεία μας, το να έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες. Και η συνθήκη τη Λισαβόνα αυτό θέλει να, να επιτύχει. Τέλο πάντων, αυτό το πρόγραμμα, γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό. Μπορεί να ακούσατε κάποιους ε, το πρωί, τον David Cameron ε, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ομιλία, στην ομιλία του στο να έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, στους πολίτες της. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Φοντάνα, τις γλωσσικές προτεραιότητες, τις ε, μειονοτικές γλώσσες, προφανώς υπάρχει, υπάρχουν τα γαλλικά στην Ιρλανδία που είναι μειονοτική γλώσσα, αλλά κερδίζει έδαφος ε, πέρα από τις καθαρά Ιρλανδόφωνες περιοχές, ε, κερδίζει πολύ έδαφος. Τώρα τα ε, γαελικά ομιλούνται σε μεγάλες πόλεις και σε όλο και μεγαλύτερο τμήμα της Ιρλανδίας. Άρα το μέλλον της γλώσσας αυτής φαίνεται μάλλον ασφαλές. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τώρα τα γαελικά είναι επίσημη, ευρωπαϊκή γλώσσα, επίσημη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα ο κόσμο στην Ιρλανδία σιγά σιγά τη μαθαίνει, τη βρίσκει, βρίσκει ότι έχει πολύ μουσικότητα και θέλει να τη μιλά όσο το δυνατόν περισσότερο. Επομένω, τα γαελικά νομίζω ότι περνάνε μια πολύ καλή περίοδο ε, στην Ιρλανδία. Όμως, ήταν μια 20 στρατηγική βάσει της οποίας ορίσαμε τις προτεραιότητές μας για τη γλώσσα μας. Γι' αυτό συμφωνώ απολύτω μαζί σας ότι η γλώσσα είναι η ταυτότητα των ανθρώπων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ολόκληρη την Ευρώπη να εξασφαλίσουμε ότι οι μειονοτικέ γλώσσε θα επιβιώσουν. Τα γαλλικά είναι μία από αυτέ τι γλώσσε. Είναι μία παλιά, αμυγό ευρωπαϊκή γλώσσα Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε το ότι θα συνεχιστεί να ομιλείτε. Έχουμε ένα πολύ ψηλό επίπεδο εκπαίδευση στην Ιρλανδία. Μερικέ φορέ ε, επικρίνουμε και του εαυτού μα. Ε, Όμω σα είπα, είχα πάει στην Κίνα, είχα μια ε, μεγάλη συζήτηση με τον Υπουργό Εκπαίδευση ε, τη Κίνα και μα είπε είναι πραγματικά πώ είναι τόσο δημιουργική η Ιρλανδία. Και του είπα ότι ο λόγο είναι ότι είναι πολύ ψηλού επίπεδου το Ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα σε ε, πολλά προγράμματα τοπικά και εθνικά η σημασία του να διαβάζει κανείς είναι πάρα πολύ, ενθαρρύνεται πάρα πολύ στα σχολεία μέσω διαφόρων προγραμμάτων, στην εκπαίδευση αλλά και εκτός ε, της εκπαίδευσης. Προς τον κύριο Κέλλη, ναι, το θέμα της δημιουργικής Ευρώπης, το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 1,8 δις είναι μικρό ποσοστό ε, της συνολικής χρηματοδότησης, είναι όμως πολύ σημαντικό. Και αν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της παγκοσμίως, πρέπει να είναι δημιουργηθεί και πρέπει να ενθαρρύνει την ε, παραγωγικότητα. Και το πρόγραμμα αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει. Γνωρίζω πολυάριθμους οργανισμούς, όχι μόνο στην Ιρλανδία, αλλά και στην Ευρώπη, γιατί είναι ευρωπαϊκό αυτό το θέμα, που αναμένουν την απόφασή μας εδώ σε σχέση με τη χρηματοδότησή μας τη μελλοντική. Γιατί πραγματικά εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση αυτή, θέλουν όχι μόνο ταχύτερη δημιουργικότητα, αλλά ξέρουν ότι δημιουργεί και θέσει απασχόληση και στο οπτικοακουστικό τομέα, αλλά και σε ολόκληρο το επιχειρηματικό φάσμα. Υπάρχουν τεράστιε συμπαραγωγέ τώρα μεταξύ χωρών ε, ε, κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρί τη χρηματοδότηση αυτή δεν μπορούν να ελοποιηθούν. Ε, ο κόσμος επίσης προγραμματίζει. Όλο και περισσότερο βλέπουν τι προγράμματα θα υπάρξουν το 2014 και όταν δεν υπάρχει σιγουριά για το πρόγραμμα αυτό και τη χρηματοδότηση θα πρέπει να καθυστερήσουν τα προγράμματά τους και το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα καθυστερήσουν και την πρόσληψη ε, προσωπικού εργαζομένων. Δεν μπορώ βέβαια να σας υποσχεθώ ότι τι, τι προϋπολογισμό θα έχουμε, αλλά αν είναι 1,8 δις, και πάλι μια αύξηση είναι. Εντάξει, είναι γεγονό ότι υπάρχουν περικοπές, λιτότητα αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω ότι είναι ένας πολύ λογικός προϋπολογισμός. Κυρία Κώστα, πραγματικά με ενθαρρύνει πολύ η συνεργασία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. και Επιτροπής. Ελπίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε πολύ καλή συμφωνία. Και συμφωνώ ότι το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο πλαίσιο αυτού πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο προπολογισμό ε, παραμένει ο μεγαλύτερο δυνατό. Να σα ευχαριστήσω λοιπόν προσωπικά για την υποστήριξή σα για το πρόγραμμα αυτό. Και όπω είπα, η διαφορά μεταξύ μας δεν είναι πολύ μεγάλη. Όταν θα υπάρξει συμφωνία στο πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία σύντομα, όλα θα πάνε καλά. Η διευκόλυνση τώρα η χρηματοδοτική είναι κάτι το καινούριο Μπορεί όμως, ε, και αυτό είναι το πιο βασικό, ε, να ενθαρρύνει τις τράπεζες ε, να βοηθήσουν την όλη διαδικασία. Είναι δύσκολο βέβαια να πάρει κανείς λεφτά από τις τράπεζες αυτή τη στιγμή, αλλά θα είναι πολύ σημαντικό για τον κλάδο αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, γιατί έτσι δίνονται κίνητρα στις τράπεζες αν όντως δανείσουν οι τράπεζες σε δημιουργικούς κλάδους, νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει κάποια σιγουριά και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Κύριε Σκούρια, έχουμε γνωριστεί στο παρελθόν ε, και έχουμε συζητήσει το πρόγραμμα αυτό. Συμφωνώ, βεβαίως, μαζί σας. Όπως και εσείς, εμείς βλέπουμε την εγγενή αξία του πολιτισμού και επίσης θέλουμε να τονίσουμε και την οικονομική αξία του πολιτισμού. Να μην ξεχνάμε ότι οι τέχνες ε, και ο πολιτισμός μεταλαμπαδεύουν το πνεύμα, ε, την ταυτότητα, την κληρονομιά ε, κάθε κοινωνίας και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τόσο μεγάλη ποικιλία ε, πολιτισμών στην Ευρώπη. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και το γεγονός ότι μπορούμε να τις συγκεντρώνουμε όλες μαζί, αυτό είναι που καθιστά αυτή τη στιγμή την Ευρώπη πολύ συναρπαστική και είναι και μια τεράστια πρόκληση για όλους μας. Είναι όμως και η ισχύ μας, είναι η δύναμή μας η δύναμή μας βρίσκεται ακριβώς στην ποικιλία αυτή. Συμφωνώ λοιπόν απολύτω μαζί σα για την αξία του πολιτισμού. Θα ήθελα ολοκληρώνοντα να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύ θετική σα ανταπόκριση. Ευχαριστώ και σας κυρία Πακ γιατί μας καλέσατε και εμένα και τον ε, κύριο Ρίνγκ ό,τι κατάλαβα από τα σχόλιά σας, πραγματικά είμαι πολύ πεπισμένος ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία πολύ καλή, πολύ επικοδομητική για το ευρύτερο καλό της κοινωνίας μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Πακ. Θα ήθελα απλώς να τονίσω, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, όπως είπατε, το πρόγραμμα για τους πολίτες είναι πολύ σημαντικό, αλλά κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί το Κοινοβούλιο δεν ακολουθεί μια κανονική διαδικασία για τον προπολογισμό. Αν το κάναμε αυτό είναι γιατί είμαστε φιλικοί προς το χρήστη, θέλουμε να αρχίσει το συντομότερο δυνατό ε, αυτό το πρόγραμμα. Ο κύριος Τάκουλα είναι εδώ που είναι σκιώδης συζητητής. Νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει και η δημοκρατική εξουσία του Κοινοβουλίου υπήρχε ένα είδο συναπόφασης, χωρίς να την αποκαλούμε βέβαια έξι, έτσι. Αν θέλετε να αποδεχθείτε τις ε, τροπολογίες μας, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία που θα βρίσκει όλους σύμφωνους και κυρίως τους ε, πελάτες. Από την άλλη, υπάρχει ο αθλητισμός. Άκουγα προσεκτικά την έκθεση για τον αθλητισμό είχα θέσει αυτό το θέμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα κάνουμε, αλλά έχουμε πολλούς περιορισμούς. Και θα χαιρόμασταν πάρα πολύ σε όλα αυτά τα διετή ζητήματα, νοστιμένων πριν του ντόπινγκ και όλα αυτά τα δυσάρεστα ζητήματα, να αρχίσουμε μια διαδικασία που θα μα βοηθήσει να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι διεθνές, αλλά πρέπει να αρχίσει με το Συμβούλιο, γιατί ο αθλητισμό δεν είναι αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου. Χαιρόμαστε όλο ιδιαίτερω να κάνουμε ακροασει το συζητάμε. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση για να σα πούμε ότι ως, ω Προεδρία, μια και σα ενδιαφέρει ο αθλητισμό, να κάνετε κάτι για αυτά τα θέματα. Από την άλλη, συμφωνώ με αυτά που είπατε σε σχέση με αυτό το διτό σύστημα, δεν μιλάω για το γερμανικό σύστημα, έτσι, μιλάω για το σύστημα που δίνει ε, στον ε, αθλητή τη δυνατότητα να έχει μια εκπαίδευση, μια κατάρτιση, να έχει τη δυνατότητα τέλος πάντων να ε, εξασφαλίσει τα προστοζήν μετά την ολοκλήρωση αθλητικής του σταδιοδρομίας. Τέλος πάντων, σας έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε. Μπορείτε και εσείς να βασιστείτε σε εμάς όταν μας λέτε τις ιδέες σας, ε, με πολύ μεγάλη χαρά θα τις ακούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να ξεκινήσουμε με τον επόμενο με το επόμενο γκρουπ υπουργών. Κύριε Φράνσις Φιτζέραλντ, Υπουργό Παιδιών και Νεολαίας και τον κύριο Κάνον, Υφυπουργό Κατάρτισης και Δεξιοτήτων που αντικαθιστά τον κύριο Ρουάρι Πιν Υπουργό Παιδείας και Δεξιοτήτων. Να σας πω καταρχάς να πω μάλλον σε κάποιους που μίλησαν για, τις μειονότητες γλώσσες. Τα Ιρλανδέζικα. Τα Ιρλανδέζικα δεν είναι μειονοτική γλώσσα. Δηλαδή είναι γλώσσα μειοψηφία, αλλά δεν είναι σε κίνδυνο υπό εξαφάνιση. Γιατί το προστατεύεται, όπως και τα Λουξεβουριέζικα Οι γλώσσες που κινδυνεύουν είναι τα κορσικάνικα, τα βρετόνικα, τέτοια. Ποιος θα ξεκινήσει? Εγώ. Κύριε Κάνον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να σας πω ότι χαίρο που μπορώ να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας μας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προς την Επιτροπή σας. Είναι τιμή που το κάνω αυτό. Ω τμήμα των, ε, της προπαρασκευαστικής δραστηριότητα, ο Υπουργό κ. Κουίν, τον οποίο εκπροσωπώ σήμερα, είχε την ευκαιρία να συναντήσει πολλούς από εσά ήδη. Συναντήσεις εξαιρετικά χρήσιμες για μας. Περιμένω, προσβλέπω σε περαιτέρω συναντήσεις μαζί σου κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Για να πετύχει οποιαδήποτε Προεδρία, πρέπει να έχει μία σχέση win-win με το Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε μια τέτοια σχέση με το Κοινοβούλιο στην Προεδρία μας. Για πολλούς στην Ευρώπη, όπως το αντιλαμβάνεστε, η κατάσταση, η περίοδος είναι δύσκολη. Οι γονεί μου ανήκαν σε μια γενιά που θέλαν τα παιδιά τους να είναι καλύτερα από αυτού. Είμαστε καλύτερα από αυτού, Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα συμβεί για τα παιδιά μα. Ω εκ τούτου, και ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης σε πολλές χώρες αυξάνεται η φτώχεια. Η ανεργία μεταξύ των νέων ιδιαίτερα έχει φτάσει καταστροφικά επίπεδα. Ο στόχος της Ιρλανδίας ως Προεδρία σε όλες τις ε, ε, εκφάνσεις του Συμβουλίου έχει στόχο να υποστηρίξει τη βιώσιμη, τις βιώσιμες θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη της Ευρώπης βασικό στοιχείο αποκατάσταση τη οικονομική σταθερότητα στην ε, ευρωπαϊκή οικονομία. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν βασικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια για την αντιμετώπιση και την επίλυση τη παρούση κρίσεω ε, ε, ανεργία στην Ευρώπη. Η ποιότητα και η δικαιοσύνη είναι οι δύο βασικά θέματα τη προεδρία μα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Και οι προτεραιότητέ μα αυτό εκφράζουν. Κάτι, οι προετοιμασίε ε, τη Προεδρία και του προγραμματό μα κράτησαν καιρό. Ο στόχο ήταν να υπάρξει συμφωνία με το Κοινοβούλιο για τα νέα προγράμματα, για το νέο πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση κατά τη νεολαία και αθλητισμό και έχουμε στόχο να ε, απαντήσουμε στην ε, έρευνα της Επιτροπής για το 2013 και για την επανεξέταση της εκπαίδευση και να συμπεριλάβουμε το ρόλο της εκπαίδευσης και της κράτηση στα πλαίσια του, της τη της Ευρώπης του 2020. Επίσης θα εξετάσουμε την κοινωνική διάσταση της ανώτερης εκπαίδευσης, την εκπαίδευση των διδασκόντων και τις δεξιότητες. Βασικός στόχος της Ιρλανδική Προεδρία στον τομέα της εκπαίδευση και τη κατάρτιση είναι να υπέρθει συμφωνία με το Κοινοβούλιο στην πρόταση για το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα στον τομέα της εκπαίδευσης κατάρτιση νεολαία και αθλητισμού. Το Μάιο πέρσι οι Υπουργοί Παιδεία τη Ένωση συμφώνησαν για μια μερική γενική προσέγγιση στην πρόταση επιτροπή. Ε, Διατηρώντα τη συνολική αρχιτεκτονική του σχεδίου κανονισμού, οι Υπουργοί πρότειναν μεταξύ άλλων να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ορατότητα ε, για την νότητα στο κείμενο με ένα χωριστό κεφάλαιο και χωριστό προπολογισμό για να εξασφαλιστεί ελάχιστη δαπάνη για κάθε τομέα του προγράμματο και να παράσχουν για μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην υλοποίηση, ιδίω σε επίπεδο εθνικών ε, γραφείων. Μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή σας 27 Νοεμβρίου πέρυσι, ξέρουμε άποψη, την άποψη του Κοινοβουλίου για την πρόταση αυτή. Η Προεδρία βάσει αυτού θα επιδιώξει εντολή από την Κορεπέρ για να, συμμετάσχει, για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την εισηγήτρια κυρία Πακ, καθώς και εκπροσώπους της Επιτροπής, εν ώψη της επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων για αυτό το σημαντικό κείμενο όσο γρηγορότερα γίνεται. Βεβαίω. Έχουμε διστάμενες απόψεις σε κάποιες από τις προτάσεις, ωστόσο σωστό είναι να πούμε ότι υπάρχει αρκετά κοινή βάση συνένεσης μεταξύ μας. Δεδομένου του κλίματος στενής συνεργασίας ε, που είχατε με την που είχαν διαφορετικές προεδρίες με την Προεδρία και με την και την ομάδα της, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε συνολική συμφωνία γρήγορα. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορούν να ξεκινήσουν έγκυρα οι προπαρασκευαστικέ δραστηριότητε για να επιτρέψουμε την θέση σε ισχύ του προγράμματο όπω προβλεπόταν την 1η Ιανουαρίου του 2014. Και αυτό θα είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά, δεδομένου του πόσο δημοφιλέ και επιτυχημένο είναι το υφιστάμενο πρόγραμμα διαβίου εκπαίδευση ναι, και, και, αλλά και του Youth in Action αλλά και άλλων προγραμμάτων, ιδιαίτερα στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε ε, χωρίς καθυστέρηση στον τομέα αυτό. Όπως ξέρετε, η ανεργία των νέων φτάνει το 23% στην Ένωση. Ταυτόχρονα, ωστόσο, υπάρχουν 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας. Η εγκατάλειψη του σχολείου νωρί παραμένει σε απαράδεκτη υψηλή, ώστε 20% των 15χρονων δεν έχουν βασικέ ικανότητε ανάγνωση. 25% των ενήλικων έχουν ε, αυτή τη στιγμή χαμηλό επίπεδο εκπαίδευση. Η Ευρώπη χρειάζεται λοιπόν να αναμορφώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα κατάρτιση και εκπαίδευση μπορούν να παράσχουν δεξιότητε και γνώσει που είναι αναγκαίε για την αγορά εργασία. Η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη λοιπόν για μα. Όπω ξέρετε, συνάδελφοι, απαντώντα στην πρόσκληση αυτή, η Επιτροπή δημοσίευσε ένα ε, ολοκληρωμένο κείμενο ανακοίνωση για την επανεξέταση τη εκπαίδευση πέρυσι τον Νοέμβριο Συμπληρωματικά με την ε, φετινή ετήσια έκθεση ανάπτυξη, η ανακοίνωση προτείνει μια σειρά προτεραιοτήτων πολιτικής για τα επόμενα έτη. Η Προεδρία μα θα είναι η πρώτη που θα απαντήσει σε αυτή τη ε, σημαντική πρωτοβουλία. Ω πρώτο βήμα η Προεδρία ετοίμασε μια σειρά συμπερασμάτων που εξετάζονται αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή εκπαίδευση εν ώψη της έγκρισης ε, στο Συμβούλιο Παιδεία του Φεβρουαρίου. Τα συμπεράσματα δίνουν νέα προκατατική απάντηση όχι μόνο στην Απροτοβουλία αλλά και στα μηνύματα που περιλαμβάνει η έκθεση τη Επιτροπή για το 2013. Η πρόκληση που έχουμε σήμερα μπροστά μα. είναι υπερβολικά μεγάλη. Δεν μπορεί να λυθεί από μία χώρα ή σε έναν τομέα. Πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε για τι σωστέ λύσει. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν για να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον. Η Ευρώπη θα πετύχει κάτι τέτοιο όταν ε, μόνο αν δώσει άτομα που έχουν και προσόντα και μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση για να συμ... και την καινοτομία. Βάσει της αιτήσης της περσινής έκθεσης για την ανάπτυξη, η έκθεση του 2013 δείχνει ότι τα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο εν ώψη τη Στρατηγική Ένωση για το 2020 για την ανάπτυξη τη εργασία. Η νέα μελέτη ρητά αναφέρει την εκπαίδευση και την κατάρτιση ω βασικέ παραμέτρου για την ανάπτυξη και την αγωνιστικότητα μαζί με την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη. Υπογραμμίζει εκ νέου το βασικό ρόλο των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο για την αντιμετώπιση της ανεργίας και για να υπάρξει μια ανάκαμψη που δημιουργεί θέσεις εργασίας υπογραμμίζοντας τη σημασία των προσόντων, της εκπαίδευσης και της διαβίου εκπαίδευσης για να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων ιδίως. Οι προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση υπογραμμίζονται και στο πακέτο Rethinking Education ε, που ανέφερα προηγουμένως. Ωστόσο ήρθε η ώρα να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε και διεξάγουμε τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδίω δε πώ χρησιμοποιούμε το έργο που έγινε με την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, ε, ε, υποστηρίζοντα τι προσπάθειε ε, σε εθνικό επίπεδο και απαντώντα τι προτεραιότητε αυτέ με ρητά, με απτά κέρδη για όλου. Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι έχουμε υπο, ε, υποβάλαμε προτάσεις για ένα στενότερο δεσμό μεταξύ των βασικών στρατηγικών προκλήσεων πολιτική που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και των δραστηριότητε που διεξήγησαν μέσω της ανοιχτή μεθόδου συντονισμού. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την στενότερη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Εκπαίδευσης και άλλων επιτροπών όπως την ε, ε, Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής και την, πολιτική, ε, και την Επιτροπή Απασχόληση. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις μεθόδους εργασίας που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της, ε, ανοιχτής μεθόδου συντονισμού για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τη συνεργασία και την γνώση από ομότιμους. Επίση θα δώσουμε έμφαση στην κοινωνική διάσταση τη εκπαίδευση, ιδίω στην ανώτερη εκπαίδευση. Χάρη στην αύξηση τη ζήτηση για ανώτερη εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια και, τις και την έλλειψη πόρων, δεν δόθηκε επαρκή προσοχή σε κάποιε σημαντικέ ανισότητε, Φερρυπίν, τα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική κοινωνικονομική ε, απόκληση. Δηλαδή τα παιδιά, των οποίων οι, φοιτητέ των οποίων οι γονείς έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευση και πόρου, έχουν μεγαλύτερε ευκαιρίε για να τελειώσουν τι σπουδέ του. Βάσει και της ατζέντα ε, για το, της Ευρώπης 2020, με στόχο να φτάσουμε το, 2020 στο 40% των 30 με ανώτερη εκπαίδευση, η Προεδρία θα προτείνει μια σειρά συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το Μάιο για την κοινωνική διάσταση της ανώτερης εκπαίδευσης. Οι αποτελεσματικέ θετικέ για την εξασφάλιση πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση σε άτομα που δεν έχουν μάθει σε σχολείο ε, που δεν έχουν διδαχθεί στο σχολείο και σε φοιτητέ ε, από, από, από, από ένα κοινωνικό background αρνητικό θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο της πρότασής μας. Φέτος, αυτό το μήνα, έχουμε και μια διάσκεψη για, την, ε, για τα ποιοτικά αποτελέσματα και την βαθμολόγηση των πανεπιστημίων. Τα 4.000 από τα 15.000 πανεπιστήμια του κόσμου βρίσκονται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να, καλεί, να, να αποτελέσει, να, παράσχει μια καλύτερη εξισορρόπηση τη σειρά των βαθμολογιών των πανεπιστημίων στον τομέα τη εκπαίδευση των διδασκόντων. Θα ασχοληθούμε με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ιδίω του εκπαιδευτού του εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί είναι βασικοί, ε, παίζουν βασικό ρόλο στην ποιότητα των σχολείων και ο στόχος είναι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να επιλέγονται σωστά και να προετοιμάζονται κατάλληλα για τα καθήκοντα που έχουν μπροστά τους. Η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών ε, είναι βασικό εργαλείο για να υπάρξει υψηλού επίπεδου διδασκαλία και καλύτερα αποτελέσματα διδασκαλίας η παροχή επαρκούς υποστήριξη στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμη για να έχουμε καινοτόμε απαντήσεις στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί. Η Προεδρία θέτει προτεραιότητα, σε αυτό το, δίνει προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό και θα προτείνει μια σειρά ε, συμπερασμάτων για την έγκριση τον Μάιο ε, στο με συμπεράσματα που θα έχουν στόχο να ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ του επαγγέλματος του εκπαιδευτή του εκπαιδευτικού, πολιτικές που θα, θα υποστηρίζουν την επιλογή τους και ανταλλαγές μεταξύ διαμορφωτών πολιτικής στους τομείς αυτούς. Εν ώψη των συμπερασμάτων θα έχουμε και μια διάσκεψη για το ρόλο του εκπαιδευτή του εκπαιδευτικού το Φεβρουάριο στο Δουβλίνο. Επίσης, θα σταθούμε στον τομέα των δεξιοτήτων θα έχουμε μια διάσκεψη το Μάρτιο που θα οργανωθεί από τη νέα υπηρεσία σε παρουσίαση προσόντων και διασφάλιση ποιότητα για τα προσόντα και την διασφάλιση ποιότητα. Η διάσκεψη αυτή θα δώσει έμφαση και στον τρόπο με τον οποίο ο χώρος της απασχόλησης και οι εμπλεκόμενοι σε αυτή χρησιμοποιούν την διασφάλιση ποιότητα για να βρουν θέσει εργασία. Κλείνοντα ευχαριστώ την κυρία Πάρκ και τα μέλη της επιτροπή, Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι θα δουλέψουμε με ρεαλιστικό και επικοδομητικό τρόπο με όλους τους εταίρου μας και θα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσει. ούτω ώστε να πετύχουμε απόδοση για όλους τους πολίτες, πραγματική απόδοση και ουσιαστική απόδοση θα μα τιμήσει πολύ αν αποφασίσετε να έρθετε στι διασκέψει μα. θα δείτε και την Ιρλανδέζικη φιλοξενία, άλλωστε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φιτσέρα τώρα. Πακ. Cumá leis an giste parlamenta seo, as ach le live anew. Is more an honor nor than féin, agus don rin lani, agus gnóhí oige. Madam Chair. I welcome the opportunity to meet the... Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω στην Επιτροπή σας σήμερα. Όλα αυτά που γίνονται, γίνονται για να εξασφαλίσουμε ότι τα 95 εκατομμύρια νέων ανθρώπων στα 27 κράτη-μέλη δεν θα γίνουν μια χαμένη γενιά. Αυτό δεν πρέπει και δεν θα γίνει. Οι προκλήσει τη παγκόσμια οικονομική κατάσταση είναι τεράστιε και αυτή τη στιγμή η παρέτηση είναι ο εχθρό μας. Η παρέτηση και η αναβολή είναι οι εχθροί μας. Το πρώτο είναι απαράδεκτο, το δεύτερο είναι αδύνατο. Είναι απαράδεκτο να παρατηθούμε και να μην αντιμετωπίσουμε τις ε, επιπλοκές της οικονομικής ε, λιτότητας και είναι αδύνατο να αναβάλουμε την ανάπτυξη, το δυναμικό, τις ελπίδες μιας γενιάς. Η εργασία των νέων είναι σημαντική για την ε, Ιρλανδική Προεδρία και για το Συμβούλιο Νεολαίας. Ο τομέα αυτός έχει να κάνει με την παροχή, με την προσφορά σε νέους ανθρώπους, ενό προγράμματος εκπαίδευση και δραστηριοτήτων, ώστε να ενισχύσουν την προσωπική και κοινωνική τους εξέλιξη. Ε, περιλαμβάνει άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση και είναι συμπληρωματική στην επίσημη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που μίλησε ο συναδελφό μου. Το ψήφισμα του Συμβουλίου για την εργασία για τους νέους το 2010 της Βελγικής Προεδρίας αναφέρει την εργασία για τους νέους ως έναν ευρύ ε, ε, όρο που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων κοινωνικής, οικονομικής, εκπαιδευτικής ή πολιτικής φύσης από, για και με τους νέους. Ε, αυτές οι δραστηριότητες βεβαίως περιλαμβάνουν και, τον αθλητισμό αλλά και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε νέους. Αυτό σημαίνει ότι η εργασία για τους νέους γίνεται εκτός ε, του, ε, της, ε, του επίσημου εκπαιδευτικού χώρου. Η, δουλειά, η εργασία για τους νέους θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νέων, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη ζωή, τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά και τις φιλοδοξίες τους. Θα πρέπει να βασίζεται στις πραγματικότητες της κάθε, του κάθε τομέα και θα πρέπει να είναι μεμονωμένοι ε, και, για να πληρεί τις ε, προϋποθέσεις ώστε οι νέοι να μπορούν να ε, βρουν τον δρόμο τους για την, για τον, για απασχόληση και για, την, για να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Βεβαίως το πρόγραμμα αυτό καλύπτει το, την πολιτική μέχρι το 2018. Περιλαμβάνει πάρα πολλές δραστηριότητε που θα γίνουν μέσω των, ε, της εργασίας για τους ε, νέους σε διάφορα κράτη-μέλη. Βεβαίως χρειάζονται μεγαλύτερη ε, γνώση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να δούμε την, ε, τις επιπτώσεις, την κλίμακα της εργασίας για τους νέους. Η Κομισιόν ε, έχει ε, ασχοληθεί με τα κενά αυτά μέσω κάποιων μελετών που έχει κάνει για την εργασία για τους νέους στα κράτη-μέλη. Αυτό θα μας βοηθήσει πολύ για να δούμε πώς είναι η κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος και θα μας βοηθήσει να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται επιτόπου στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι σημαντικό γιατί τα κράτη-μέλη ε, ε, επενδύουν σημαντικά σε τέτοιες δραστηριότητε. Είναι όμως δύσκολο προς το παρόν να ε, αξιολογήσουμε την, την κλίμακα ε, αυτών των δραστηριοτήτων ε, λόγω του τρόπου ε, χρηματοδότησης και οργάνωσης αυτών των δραστηριοτήτων σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Πολλές δραστηριότητες μπορούν να, γίνουν, να χρηματοδοτηθούν από σπόνσορες στα κράτη-μέλη, αλλά και οι εθελοντές συμβάλλουν πολύ σημαντικά. Σε άλλα κράτη περισσότερο, σε άλλα λιγότερο. Σημαντικό όμως είναι να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη δέσμευση σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας, σε όλα τα κράτη-μέλη, για τις επενδύσεις που θα είναι αποτελεσματικές για τους νέους ανθρώπους. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν όντω λειτουργεί η εργασία για του νέου και αν μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Αυτό θέλουμε να ε, ε, εξερευνήσουμε και σε αυτό θέλουμε να καταλήξουμε στα συμπεράσματά μα. Με τη βοήθεια βεβαίω και των νέων ε, από τα κράτη-μέλη. Ε, οι πρόσφατε εξελίξει στην πολιτική λένε ότι η εργασία για του νέου ε, περιέχει δυναμικό ώστε να γίνουν περισσότερα και κυρίω αφορά του νέου που ήδη βρίσκονται περιθωριοποιημένοι από την εκπαίδευση, από την κατάρτιση, από την εργασία, από την απασχόληση. Όλε οι εκθέσει που σα ανέφερα και η Ευρώπη 2020 αναγνωρίζουν ακριβώ το δυναμικό που έχει η εργασία για του νέου ώστε να καλύψει τι ανάγκε αυτή τη ομάδα νέων. Ξέρουμε ότι η κρίση στην Ευρώπη έχει ε, σημαντικέ επιπτώσει, δεν χρειάζεται να πω εγώ πολλά. σημαντικές επιπτώσεις για τους νέους. Το πρόβλημα τη της, ε, ε, ε ανεργία των νέων είναι σημαντικό. Η αύξηση είναι εξαιρετική σε σχέση με, την, ε, ε σε σχέση με, το, με τις ηλικιακές ομάδες που πλήττει. Από 15 24 ετών έχουμε αύξηση 50%. Και αυτό κυρίω αφορά άτομα που δεν βρίσκονται σε ένα επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον. Και αυτό σημαίνει ότι περίπου 7,5 εκατομμύρια νέων ανθρώπων ε, μεταξύ 15 και 24 ετών βρίσκονται σε πολύ ψηλό κίνδυνο φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού και βεβαίως ξέρουμε ότι αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο της, απειλέ τις απειλές για την υγεία αλλά και για την ευημερία τους. Το Eurofund έχει κάνει κάποιες ε, μελέτες ε, και δείχνουν ότι υπάρχει τεράστια οικονομική απώλεια περίπου 153 δισεκατομμυρίων σε ό,τι αφορά την οικονομική και, το, τις οικονομικές και κοινωνικές απώλειες λόγω του ότι αυτοί οι νέοι δεν συμμετέχουν στους κλάδους που σας ανέφερα και δεν έχουν τις ευκαιρίες που χρειάζονται ώστε να συμμετέχουν αυτό μπορεί να ε, μετρηθεί. Αλλά υπάρχουν πολλά που δεν μπορούν να μετρηθούν σε σχέση με αυτές τις προκλήσεις. Ε, το, αυτό, ας πούμε, το, αυτό που δεν μπορεί να μετρηθεί είναι ε, ακριβώς η μη συμμετοχή του στην κοινωνία. Είναι διαβροτική λοιπόν αυτή η, αυτή η, απουσία τους από την ε, από την αγορά εργασία, ε, προφανώ μειώνει τι δυνατότητε του ε, για δημιουργικότητα, για καινοτομία, για επιχειρηματικότητα και για προσαρμοστικότητα, ε, Αρετέ που είναι πραγματικά πολύ χρήσιμε ώστε να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική ευημερία στα κράτη-μέλη. Η Προεδρία λοιπόν θέλει να μετρήσει το δυναμικό και να αξιοποιήσει το δυναμικό των υπηρεσιών που ασχολούνται με την εργασία των νέων, έχοντα βεβαίω και την υποστήριξη των, ε, ε, των ε, δικτύων των νέων. Βεβαίως προσβλέπουμε με το τρίο των Προεδριών, την Λιθουανία και την Ελλάδα, που έχουμε κάνει πολύ σημαντικές συζητήσεις για τα προγράμματα κοινωνικής ε, ένταξης να προωθήσουμε τις προτεραιότητες ε, της ε, Προεδρίας μας. Να εξερευνήσουμε δηλαδή το δυναμικό της εργασίας για τους νέους και των δραστηριοτήτων για τους νέους, ειδικά στα πλαίσια του Ευρώπη 2020, να προωθήσουμε την κατανόηση της ποιοτική εργασίας για τους νέους και πώς μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των νέων στην κοινωνική του συμπερίληψη και να ολοκληρώσουμε τον πρώτο κύκλο διαλόγων μεταξύ νέων και ε, χαρασόντων πολιτική. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο της δουλειάς μας. Μεταξύ και του Συμβουλίου και του Κοινωνιβουλίου και τη Κομισιόν, μαζί με του νέου θα συνεργαστούμε για να τα καταφέρουμε. Θα εργαστώ βεβαίω εγώ από κοινού με τον ε, Υπουργό Εκπαίδευση υπάρχει και η δική σας ε, έκθεση που, αφορά ένα, που έχει ένα κεφάλαιο αποκλειστικά για, την, για τους νέους. Ε, και έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε και του στόχου του Ευρώπη 2020. Πρέπει να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες συμμαχίε και σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο για όλους αυτούς τους τομείς, όπω η νεολαία, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η απασχόληση. Όπως είπα, η Ευρώπη 2020 έχει να κάνει και με την κοινωνική Ευρώπη. Η πολιτική για την εργασία των νέων έχει να κάνει και με πολιτικά και με κοινωνικά θέματα και όχι μόνο με οικονομικά. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση γίνεται συχνά εκτός ε, σχολείων, ε, όχι μόνο σε παραδοσιακές εγκαταστάσεις. Ε, δουλεύει για τους νέους με το δικό τους ρυθμό γιατί θέλουν να συμμετέχουν. Κάνει αυτό το οποίο κάποια πιο επίσημη αντίδραση δεν μπορεί να κάνει. Ε, είναι πάνω από συμπληρωματική στην επίσημη εκπαίδευση, κατάρτιση. Ε, δίνει βέβαια περισσότερη αξία, ε, αξία που δεν μπορεί να υπολογιστεί βέβαια. Μία πολιτική για τη νεολαία συντονισμένη με άλλους τομείς σχετικούς θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στα, στην υγεία, στην ευημερία, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην απασχόληση των νέων και πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ ανθρώπους, τους νέους που έχουν ε, πρόβλημα ε, συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Ε, το Συμβούλιο των Νέων το Μάιο του 2013 θα κληθεί να δώσει συστάσεις εν ώψη της πολιτικής νεολαίας ε, στην Ευρώπη 2020 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα ενημερωθούν από, το, από την διάσκεψη των νέων για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα γίνει το Μάρτιο στο, Δουβλίνο. Υπάρχει μια, ένας διαδρομένος διάλογος με τους νέους στην Ιρλανδία. Είναι μια διαδικασία την οποία πραγματικά την υποστηρίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί ε, η άποψη των νέων ε, και βλέπουμε όλο και περισσότερο την άμεση δέσμευση και συμμετοχή ε, της νεολαίας στην ανάπτυξη των πολιτικών και αυτό φυσικά είναι κάτι πρέπει να το επικροτούμε. Επίσης θα γίνει και ένας νέος γύρος τραπέζης τον Ιούνιο στο Δουβλίνο με τους νέους και όπως είπε και ο συνάδελφος αναμένουμε εναγωνίως την συμμετοχή των μελών ε, της Επιτροπής σας. Ε, επίσης θα ήθελα να πω ότι μπορεί να μπορούμε να μετρήσουμε τις άμεσες συνέπειες ε, του γεγονότος ότι μια γενεά νέων ανθρώπων απομακρύνονται από την κοινωνία και απογοητεύονται. Πρέπει να μπορούμε όμως να δούμε την ποιότητα, να μετρήσουμε την ποιότητα Τη ε, εργασία των νέων. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να την ενθαρρύνουμε. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανώσει των νέων ε, ε, θα πρέπει να ε, έχουν ε, αποτελεσματικά προγράμματα προς όφελος των νέων, ε, να λαμβάνονται υπόψη οι εμπειρίες τους, οι απόψεις τους και επίσης πρέπει να εστιάσουμε στα αποδεικτικά στοιχεία, στα αποτελέσματα. Όλο και περισσότερη έρευνα εθνική και διεθνής μας λέει τι είναι αποτελεσματικό στη συνεργασία μας με τους νέους. Όπως έχουμε περισσότερα ερευνητικά στοιχεία σε σχέση με προηγούμενες προσπάθειες. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο περισσότερα για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να διευκολύνουμε τους νέους. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όφελος από τη συμμετοχή. Αν οι, άνθρωποι, αν οι νέοι θέλουν να συμμετέχουν σε εργασία για την νεολαία, πρέπει να τους δώσουμε και ένα μέγιστο όφελος. Ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό που έμαθαν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και της ζωής τους και να αναγνωρίζεται αυτό. Ε, η οργάνωση της δουλειάς αυτής ε, είναι διαφορετική σε κάθε κράτος μέλος ε, και αυτός ο πλούτος είναι πολύ απαραίτητος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες διαστάσεις των αναγκών και των εμπειριών των νέων. Ε, δι, βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη προδιαγραφών ποιότητα στα κράτη-μέλη και θα ξεκολουθήσουμε να την ενθαρρύνουμε κατά τη διάρκεια τη Ιρλανδική Προεδρία. Επίση, ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε την κοινή κατανόηση τη ποιότητα τη δουλειά για του νέου και την ύπαρξη προδιαγραφών στι δραστηριότητε των νέων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι η Επιτροπή σα ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ανάπτυξη των προδιαγραφών όπω κάνατε και στην διαβίου εκμάθηση και επίση θα παρακολουθήσουμε συστηματική συστάσεις και προτάσεις ε, που ε, θα υπάρξουν για την ε, κινητικότητα των νέων, για την κάρτα κινητικότητας των νέων δεν ε, υπάρχει τίποτε που να αφορά τους νέους χωρίς τη συμμετοχή τους. Αυτό είναι μια βασική αρχή και είναι ένα βασικό στοιχείο της δουλειάς ε, την οποία σας παρουσίασα. Ε, ελπίζω να έχουμε πολλές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας να προωθήσουμε αυτές τις προσπάθειες με τη δική σας, με συνεργασία και έχουμε επίσης και μια ανεπίσημη συνάντηση υπουργών αρμοδίων για τα θέματα αυτά στο Δουβλίνο και θα έχουμε και ένα διαδρομένο διάλογο για... και θα έχουμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα κάνουν τη διαφορά. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε επίσης ότι έχουμε την εμπειρία που έχουμε ε, στην αξιοποίηση της εμπειρίας των νέων και θέλουμε να έχουμε ένα θετικό αντίκτυπο στη ε, ζωή των νέων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να παρουσιάσω τα σχέδια της Ελληνικής Προεδρίας και με πολύ χαρά θα συνεργαστώ μαζί σας για τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στη συζήτηση, λέει η Πρόεδρος. Να δώσω το λόγο στον κύριο Πέκερ που ε, ήθελε από πριν ήδη να θέσει ένα ζήτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε ο κύριος Κάνον, η διαβίου μάθηση είναι στον πυρήνα των ε, δραστηριοτήτων της Προεδρίας. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό και ε, από την οπτική γωνία τούτη τη Επιτροπή θα ήθελα να τονίσουμε ότι έχουμε ε, συμβάλει πολύ έτσι ώστε να υπάρχει ένα εξαιρετικό ε, προϊόν τελικά. Μιλούμε για το μέλλον αυτής της γενιάς και αυτός είναι ένας από τους πυλώνες για την αντιμετώπιση των εχθρικών πεπιθήσεων απέναντι στην Ευρώπη. Και βεβαίω η αντιμετώπιση τη ανεργία των νέων είναι σημαντικό θέμα. Αυτό που περιμένουμε από εσά είναι να μα να μας στηρίξετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Δεν μπορούμε να, υπάρχει, να, να έχουμε εδώ ε, πολιτικέ λιτότητα, γιατί ακριβώ έτσι ε, θα, δεν θα επιτύχουμε τους στόχους που θέλουμε. Δεύτερον, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την, ε, την κυρία Φιτζέραλτ για, όσα, για τα όσα είπε, για την εργασία των νέων. Είναι πολύ ενδιαφέρον το μοντέλο που μας παρουσίασε και θέλει όντως να ε, χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό που υπάρχει. θα ήταν καλό να υπάρχει ένα μοντέλο των πρακτικών. Ξέρετε ότι υπάρχει και η επαγγελματική κατάρτιση που στα κράτη-μέλη ε, πολλές φορές έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Και το δικό μου αίτημα προς εσάς, η δική μου έκκληση, είναι αυτό το benchmark να το χρησιμοποιήσετε, να το μελετήσετε, γιατί αυτές οι χώρες και τα ε, ε, ιδρύματα που το προσθέτουν είναι σε θέση και να συμμετέχουν στον διάλογο ενεργά, γιατί εδώ μιλούμε όχι για λεφτά, μιλούμε για ταχύτητα. Γιατί οι διπλή, ε, τα συστήματα διπλής ε, εκπαίδευσης χρειάζονται χρόνο και ε, θα πρέπει εδώ αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Γιατί αυτές οι έννοιες υπάρχουν, δεν χρειάζεται να τις εφεύρουμε, αλλά η εφαρμογή τους, εκεί ακριβώς χρειάζεται μια έξυπνη προσέγγιση. Και ελπίζω να το κάνετε αυτό κατά τη διάρκεια της προεδρίας. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Λόκεγκάρντ έχει το λόγο. Thanks, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους Υπουργούς ε, για την ε, δέσμευσή τους ε, και την καλή και σαφή παρουσίασή τους. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτό που είπε ο κύριος Μπέκερ σε σχέση με το θέμα των χρημάτων. Καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία σήμερα ούτε μια θέση από πλευρά Συμβουλίου γιατί είμαστε ακόμη σε διαπραγματεύσει, Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μήπω θα μπορούσατε να μας πείτε κάποιο είδους, να μας δώσετε κάποια είδου ένδειξη. Μιλάμε για διατήρηση του status quo ή αύξηση, γιατί και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποστηρίζουμε μία αύξηση 17% ε, σε αυτό το ε, εξαιρετικό πρόγραμμα, κάποιο είδους ένδειξη θα μας ήταν πολύ χρήσιμη. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα το ίδιο να πω, γιατί έχουμε πολλές φορές αναφέρει πόσο σημαντικό είναι, ε, είναι σημαντική η, εκπαίδευση, η κατάρτιση για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ειδικότερα όταν πρόκειται, από τους, όταν για τους νέους, για να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας για ένα καλύτερο μέλλον και για να αντιμετωπίσουμε και την ανεργία. Ξέρουμε ότι έχουμε μια μάχη για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί υπάρχουν τάση στο Συμβούλιο ότι θα υπάρξουν οι παλαιότερες ε, προτεραιότητες, διαφορετικά ταμεία δηλαδή και γεωργία κατά παραδοσιακό τρόπο. Ε, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός, ε, η αύξηση του προϋπολογισμού που ζητούμε εμείς για την έρευνα, την νεολαία, την εκπαίδευση και τις σχετικές δραστηριότητες θα μειωθούν θα μειωθεί. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας, ε, ποια είναι η άποψή σας ε, σε σχέση με τον αγώνα αυτό που πρέπει να δοθεί και για τα προβλήματα με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτη ερώτηση προς τον Υπουργό. Τονίσατε την προσαρμοστικότητα, την, τη δυνατότητα προσαρμογής του φοιτητή, του μαθητή στην θέση εργασία. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Ο κόσμος αλλάζει. Σήμερα μια δουλειά καλή είναι απειρχαιωμένη, είναι παραγωνισμένη σε λίγα χρόνια. Πέραν της επαγγελματικής και προσαρμόσιμης κατάστασης, κατάρτισης, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια βάση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψει την μελλοντική προσαρμογή δεν πρέπει να, προς, ε, να προσανατολιζόμαστε υπερβολικά στην, ε, στον, στην έβρεση ε, θέσεων εργασίας σήμερα. Μιλήσατε για τα ranking των πανεπιστημίων, τη βαθμολόγηση των πανεπιστημίων. Τι εννοείτε, μπορεί να λειτουργήσει, θα δημιουργήσετε μια νέα μορφή ε, ε βαθμολόγησης, γιατί το υφιστάμενα συστήματα δίνουν κακή βαθμολογία στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μπορείτε να μας πείτε επίσης τι συστάσεις έχετε στη μάχη κατά της εγκατάλειψης του σχολείου. Πανεπιστήμια. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία κοινωνική αναπαραγωγή. Δηλαδή, οι νέοι που φτάνουν σε ψηλέ θέσει στο πανεπιστήμιο έχουν γονείς που έχουν κάνει σπουδές. Αυτό σημαίνει ότι το κοινωνικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Τι συστάσεις έχετε για να λύθει το ζήτημα της, του κοινωνικού της κοινωνικής διάστασης του πανεπιστημίου σκέφτες, για παράδειγμα, το ενδεχόμενο να υπάρχει ένα επίδομα στέγης. Συχνά τα πανεπιστήμια είναι σε μεγάλες πόλεις και είναι δύσκολο να βρει ο φοιτητή ε, στέγη. Τι συστάσεις έχετε για τους φοιτητέ που προέρχονται από λαϊκά στρώματα. Θέλω να τονίσω επίσης το εξής. Τι θα κάνετε για να για στη μάχη του προπολογισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είπατε πολλά πράγματα. Αν δεν υπάρχουν χρήματα ωστόσο, θα είναι ωραία λόγια και θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της αξιοπιστίας της Ένωσης, ιδίω για τους νέους. Κύριε Φιτζέραλντ, εκτιμώ ιδιαίτερα την εικόνα που παρουσιάσετε, είναι ενδιαφέρουσα, την υποστηρίζω. Μιλήσατε για τον κίνδυνο να έχουμε 95 εκατομμύρια νέων που θα αποτελέσουν μια χαμένη γενιά χωρίς δουλειά, χωρίς ένταξη. Πώς βλέπετε την ανάπτυξη της αυτονομίας των νέων. Μιλήσαμε, μιλήσατε για μια εγγύηση για την νεότητα. Είναι σύσταση αυτή, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα το προχωρήσετε. Θα χτυπήσετε, θα ζητήσετε από τα κράτη-μέλη αυτή η εγγύηση για τους νέους να μην είναι ευχολόγιο, αλλά να υλοποιηθεί πραγματικά από τα κράτη-μέλη. Αλλιώς θα έχουμε μια χαμένη γενιά νέων χωρίς δυνατότητα αξιοπρεπούς ζωής. Μιλήσατε για έναν κύκλο διαπραγματεύσεων μεταξύ νέων και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων. Τι ημερήσια διάταξη θα υπάρχει, τι θέματα θα συζητηθούν. Euh, για τη σπουδαιότητα της αναγνώρισης των προσόντων το αναφέρατε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μιλήσατε για την υποστήριξη μιας ομάδας εθελοντών νέων που μπορούν να δουλέψουν ε, χωρίς ε, μισθωτή εργασία αναγκαστικά, κάτι που είναι περίπλοκο. Δουλεύετε για αυτή την προσέγγιση της εθελοντικής δουλειάς, με ποια με, ποια, με ποιο σκεπτικό. Θα αλλάξετε τον κόσμο, βλέπω, ε. Τέλος πάντων. Κύριε Κέλλη, σύντομα αν θέλετε. Indeed, Madam Chair. Ε, Μάλιστα. Καταρχάς, να καλωσορίσω τους δύο υπουργού. Η κυρία Φιτσέραλντ είναι η πρώτη υπουργός ε, νέων στην ιστορία της χώρας μας ε, και χαίρομαι που έγινε το δημοσχετικό δημοψήφισμα για την εξασφάλιση των δικαιώματων των παιδιών. Ένα ερώτημα ήθελα να θέσω ε, για το πρόγραμμα εγγυήσεων. Είναι ικανοποιημένη η Υπουργός. Είναι θέμα κλειδί για τους νέους ώστε να μπορέσουν να έχουν θέσεις εργασίας. Για τον κύριο Κάνον. Το καλοκαίρι για έναν φιλανθρωπικό σκοπό κάναμε έναν αγώνα ποδηλατο, ποδηλατοδρομία ε, και τελειώσαμε και δύο βεβαίω. Φτάσαμε στο τέρμα, ευτυχώ. Ε, μιλήσατε για την εκπαίδευση, την κατάρτιση. Με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό που είπατε για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και το πώ μπορούμε να, να, να, να αυξήσουμε το δικό του επίπεδο σε όλη τη διάρκεια τη καριέρα του. Πώ μπορεί να γίνει αυτό, Έχετε αποφασίσει για κάποια θέματα πόσο συχνά θα γίνεται κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Τάκουλα δεν είναι εδώ. Η κυρία Σάντσες Σμίτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε και κυρία Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πίστη σας και την ενέργεια και τη βούλησή σας να αφιερωθείτε σε αυτή την Προεδρία που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική για μας γιατί το 2013 είναι εξαιρετική σημασία. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι εκφράσεις που χρησιμοποιήσατε, ο διάλογος με την νεολαία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η νέα η νεολαία να αισθάνεται ότι θα μπορέσει να διαμορφώσει το μέλλον της, ότι πράγματι η παρέτηση δεν θα πρέπει να αποτελεί τμήμα του λεξιλογίου μας. Όλοι είμαστε πεπισμένοι για τη σημασία της ε, εκπαίδευσης, της κατάρτισης. Η στρατηγική 2020 επιζητά ευφυή ανάπτυξη μας λέτε να βελτιώσουμε αυτά που υπάρχουν και μιλάω για το νέρασμο που αποτελεί, ήταν αντικείμενο μεγάλων συζητήσεων ε, και δεν μιλάω μόνο για το ότι αποκαλείται έρασμος, μιλάω για οτιδήποτε ε, αφορά κινητικότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό η πρόσβαση για την ε, στην... ενημέρωση, στην κατάρτιση συγγνώμη, για όλους, γιατί έχει άμεση σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση. Και το λέω αυτό γιατί θέλουμε επίσης να προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας και στην αγορά εργασία στην ανώτερη εκπαίδευση. Δεν έχει νόημα δηλαδή μόνο να προσφέρουμε, ε, να προσφέρουμε ε, ε, εργαζομένους στις επιχειρήσεις. Οι νέοι μας πρέπει να είναι σε θέση να διαλέξουν το μέλλον τους. Μα δώσατε ήδη κάποιε απαντήσει, αλλά δεν θα ήθελα να μα διαφεύγει ότι υπάρχουν και άλλα ε, ταμεία που μπορούν να μα βοηθήσουν στι προσπάθειε μα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για παράδειγμα, να μην ξεχνάμε και τα περιφερειακά ε, ταμεία, τα οποία επίσης μπορούν επιτόπου να μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Και το θέμα της διευκόλυνσης για την νεολαία που ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια, Ελπίζω να γίνει μια πραγματική πρωτοβουλία και να μην παραμείνει απλώς ένα ψήφισμα και μια ε, ε, επιθυμία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καμεβέρτη. Ευχαριστώ. Σύντομα. Καταρχά να ευχαριστήσω τους υπουργού για, ε, για τις παρεμβάσεις τους. Κυρία Φιτζέραλτ, χαίρομαι που αναφέρατε την σημασία της άτυπης εκπαίδευσης, κυρίως για τους νέους και ότι προφανώς είστε διατεθειμένοι να υποστηρίξετε την προσέγγιση μας εδώ στην Επιτροπή για να υπάρχει ένα κεφάλαιο ειδικά για τους νέους στο νέο πρόγραμμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, το έχουμε πει, ότι ακριβώς το θέμα της άτυπη εκπαίδευση είναι τόσο ε, ολοκληρωμένος τομέας που θέλουμε να διατηρηθεί ε, ξεχωριστά. Πάντα μιλούμε για τη στρατηγική 2020 είναι σημαντική. Βλέπουμε όμως όλοι ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων είναι μία από τις βασικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε προς το παρόν και αυτό πρέπει να το λύσουμε άμεσα. Πάντα με, με φοβίζει εμένα όταν αυτό το αναφέρουμε σε σχέση με τα προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία συζητούμε εδώ στην Επιτροπή. Γιατί πάντα μου δημιουργείται ανησυχία ότι δημιουργούμε λάθος εντυμός, εντυπώσεις και δημιουργούμε ψευδείς προσδοκίες. Αυτά που κάνουμε με τούτα, τα λίγα λεφτά και με τα προγράμματα που έχουμε είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά για μας, είναι πολύ σημαντικά ε, αλλά το να δημιουργούμε την, ε, την εντύπωση ότι με αυτά τα προβλήματα μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της ενεργείας των ε, νέων και της εκπαίδευσης εν γέννη, προφανώς αυτό θα είναι μοιραίο για μας. Χρειαζόμαστε άλλα εργαλεία. Ο κύριος Μπέκερ μίλησε για τα συστήματα διπλής εκπαίδευσης. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, νέε ιδέε. Χρειαζόμαστε τα διευθυντικά ταμεία. Γιατί, εντάξει, πάλι για λεφτά λέω, αλλά έχει να κάνει και με το πόσα χρήματα έχουμε και πόσα, μπορούμε να, πόσα προγράμματα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και στην εκπαίδευση και στη μετεκπαίδευση των, νέων, των νέων. Αυτά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνο με τα δικά μας ε, προγράμματα. Μιλούμε για κινητικότητα, μιλούμε για την, για το να θέσουμε τους νέους στο επίκεντρο των προγραμμάτων για να αξιολογήσουμε, για να εκμεταλλευτούμε ακριβώς το ανθρώπινο κεφάλαιο, για να μπορέσουμε όλα αυτά να τα προωθήσουμε και να φέρουμε και την Ευρώπη ένα βήμα πιο μπροστά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά θα πρέπει πάντα να τα τονίζουμε, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπωσει. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Κάνον ή η κυρία Φιτσέρολ θα πάρει πρώτα το λόγο. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Εσείς. Παρακαλώ. Um, ε, ευχαριστώ πολύ. Υπήρξαν πολλέ ερωτήσει που είχαν να κάνουν με τον έρασμο και νομίζω ότι ο συνάδελφο ε, θα τι απαντήσει λεπτομερέστερα γιατί είναι η δική του αρμοδιότητα κατά βάση. Ε, εγώ αναφέρθηκα βέβαια στη σημασία των ταμείων, τη σημασία της εκμάθησης και των διαφόρων ευκαιριών που μπορεί να υπάρξουν. Κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω συμβατότητα σε αυτό που είπατε σε σχέση με τις ροές ε, χρηματοδότησης ε, και την ε, ανεπίσημη εκμάθηση. τη σημασία το να θεωρείται όχι μια μεταβατική περίοδος απλώς προς την απασχόληση, αλλά να θεωρείται μια σημαντική αυτόνομη περίοδος στη ζωή των νέων η εκπαίδευση και η εκμάθηση πρέπει να υπάρχουν πρέπει να, να υπάρξει ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε και άλλα ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για τους νέους σε σχέση με την απασχόληση, τις δεξιότητες ε, ε, όπως η αυτοπεποίθηση, το ηγετικό πνεύμα και όλα αυτά θα έχουν αντίκτυπο και σε, άλλες, σε άλλους τομείς. Αλλά καταλαβαίνω, είναι σημαντικό ε, να υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια Επίσης, ε, αυτό που είπατε σε σχέση με το κεφάλαιο ε, στην αγορά δεν αφορά φυσικά μόνο αυτό. Ε, υπάρχει και το θέμα της ασυμβατότητας με την αγορά εργασίας. Για το ερώτημα του κυρίου Μπέκερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και θα ήθελα να σας, να σας διαβεβαιώσω ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τα ε, αποτελέσματα σε σχέση με την κατάρτιση και την εκπαίδευση είναι η αναγνώριση ότι υπάρχει καλή πρακτική, ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις ε, καλύτερες πρακτικές από τα κράτη-μέλη, να αξιοποιούμε ε, τις καλύτερες πρακτικές. Είπατε ότι υπάρχουν πολλά μοντέλα όντω και πρέπει κάπως να τα συγκεράσουμε για να υπάρξει εφαρμογή. Δεν αφορά δηλαδή μόνο την ε, συγκέντρωση των μοντέλων, πρέπει να εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη, να εξασφαλίζουμε ότι θα... Ε, εφαρμόζονται και να βλέπουμε και τις βέλτιστες πρακτικές. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές, αυτό το γνωρίζω. Ε, δεν είναι δυνατόν κανείς να επιβάλλει μια προδιαγραφή από πάνω προς τα κάτω. Πρέπει να δει τι γίνεται, να πει υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές, ότι πρέπει να τις συγκεντρώσουμε και να υπάρχει ένα ε, πλαίσιο ε, ποιοτικό μόνο πάνω από το οποίο θα, θα, θέλουμε να πάμε. Είναι σημαντικό το θέμα του προϋπολογισμού. Ε, Ιρλανδική Προεδρία το γνωρίζουμε αυτό, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπάρξει εστίαση ε, σε αυτά τα θέματα. Πολλοί ευρωβουλευτέ το έθεσαν, το θέμα της κοινωνικής Ευρώπης και τη σημασία των προγραμμάτων αυτών για του πολίτε και την κατανόηση ε, της Ευρώπης ε, από του πολίτε, Θα συμφωνήσω βεβαίω με αυτό και όταν είμαι στο Δουβλίνο και με τους επιτρόπους έχω πολύ ε, έντονες συζητήσεις σε σχέση με ε, το θέμα αυτό δεδομένου, δεδομένης οικονομικής συγκυρίας. Πρέπει να επικεντρωθούμε βέβαια και στις οικονομικές πτυχές αλλά και στις κοινωνικές ε, πτυχές που είναι κεφαλαιόδου σημασίας για τους πολίτες μας. Γιατί πρέπει να έχουμε μια θετική και πολύτιμη συνεισφορά στη ζωή των συμπολιτών μας. Ε, ένας ε, συνάδελφος επίσης μίλησε για τις νέες δυνατότητες για τα παιδιά, ε, να μην πάμε δηλαδή απλώς στις παλαιότερες προτεραιότητες, παλαιότερες προτεραιότητες αλλά να τονίζουμε και τις προτεραιότητες που η Επιτροπή σας εντόπισε. Φυσικά αυτό έχει ήδη οριμάσει ως σκέψη στην Ιρλανδική Προεδρία και νομίζω ότι την τελευταία, την περασμένη εβδομάδα που μίλησε στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, το είπα αυτό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια κοινωνία καλή για τα παιδιά μα, να μεγαλώσουν σε μια καλή κοινωνία, να συναλλάσσονται επιχειρηματικά σε αυτή την ε, ε, ε, κοινωνία, να γεράσουν σε αυτή την κοινωνία με την αντίστοιχη υποστήριξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για να το πετύχουμε πρέπει νωρί να επενδύσουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ο Ευρωβουλευτής Κέλλη, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας καταρχάς. Ε, Σον, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ε, εγγύησης για τους νέους. Το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ε, νομίζω ότι και ε, συνάδελφός μου σε άλλη επιτροπή το έθεσε αυτό το ζήτημα και έδωσε ιδιαίτερες ιδιαίτερη προτεραιότητα στην πρόοδο σε σχέση με τις συστάσεις για την εγγύηση αυτή για την νεολαία ε, και επίσης θα το θέσουμε και στο, στη συνάντηση ΕΠΣΚΟ στο τέλος του ε, Φλεβάρι. Θα συνεργαστούμε ε, με τη συνάδελφο την αρμόδια για να εξασφαλίσουμε ότι όντως θα προωθήσουμε αυτό το ζήτημα. Ε, κυρία Σμιτ, μιλήσατε για το διάλογο με τους νέους. Ναι, όντω ε, γίνεται αυτό ο διάλογο. Υπήρξε και ερώτημα προηγουμένω για αυτό το θέμα από άλλο συναδελφό σα σε σχέση με το πότε θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα αυτού του διάλογου. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει του τελευταίους μήνες. Έχει δρομολογηθεί και στα κρατη κατά, κατά τον τελευταίο χρόνο. Χιλιάδες νέοι ε, ήταν, ε, συμμετείχαν στη διαβούλευση. η έκβαση θα γνωστοποιηθεί στη διάσκεψη με τους νέους το Μάρτιο. Αλλά πέρα από αυτό, σε κάθε κράτος μέλος υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για να ακουστεί η άποψη των νέων ε, ανθρώπων, ε, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που συμμετείχαν σε ε, εργασία για τους νέους, στα σχολεία. Ε, σημειώνουμε πολύ μεγάλη πρόοδο σε σχέση με τη συνεργασία με τους νέους. Είναι μια πραγματικότητα επιτόπου. Δεν το λέω απλώς. Ναι, γίνεται όντως στην, στην καθημερινή ζωή και Πραγματικά είναι πολύ χρήσιμη η ζωτικότητα και η ενέργεια των νέων. Είναι σημαντικό να ακούσουμε την άποψή τους για να ξέρουμε τι κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε στις πολιτικές μας. Νομίζω αυτά. Ευχαριστώ. να σχολιάσω δύο-τρία πράγματα που αναφέρθηκαν επανειλημμένα σε, όλα τα, σε όλες τις παρεμβάσεις. Μιλήσατε για τον προϋπολογισμό οι περισσότεροι. Εμεί υποστηρίζουμε έναν προπολογισμό ο οποίο θέλει να, ενισχύσει την ε, δημιουργία θέσεων εργασία και, την ανάπτυξη και κυρίω την, ε, το θέμα τη θέση εργασίας, θέσεων εργασία. Δηλαδή να υπάρχουν και άνθρωποι που θα καλύψουν αυτέ τι θέσει εργασία όταν αυτέ θα προκύψουν. Πρέπει λοιπόν να το δούμε γιατί αυτό ο τομέα είναι ένα τομέα που μπορεί να βοηθήσει. και θα ενισχύσουμε βεβαίω και τα κρατημέλη και του εταίρου μα, ε, όσο μπορούμε. Ο πρόεδρο Φαν είπε ότι πρέπει να υπάρξει σύγκληση για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το πολυετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα το δούμε βεβαίως αυτό και το Φλεβάρι. Η διαβίου μάθηση επίσης είναι ένα σημαντικό εργαλείο, ένα από τα εργαλεία που μπορούμε να βοηθήσουμε τους ε, πολίτες μας να επανέλθουν στον χώρο εργασίας. Ετέθη το θέμα και της απομάκρυνσης από τις παραδοσιακές μεθόδους και αυτό το υποστηρίζω. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει δραστικά Ίσως λοιπόν και τα ε, συστήματα εκπαίδευσης να μην κινούνται με την ίδια ταχύτητα. Μέχρι το 2025 50% των, ε, της, ε, των επαγγελμάτων που θα υπάρχουν δεν, θα δεν υπάρχουν σήμερα και δεν έχουμε λέξεις να τα περιγράψουμε. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μείνουμε πίσω στα συστήματα εκπαίδευσή μα. Ότι αυτή η καινοτομία που υπάρχει στον κόσμο, τη τεχνολογία κυρίω, θα μπορέσουμε να την παρακολουθήσουμε. Μιλήσατε για, τα, για τις δεξιότητες, όχι μόνο τις ακαδημαϊκές. Αυτό είναι όντως ένα από τα σημεία στα οποία θα επικεντρωθεί η Προεδρία μας, κυρίως στα πλαίσια της διαβίου μάθησης. Γιατί όντω θέλουμε οι νέοι μα να έχουν τι δεξιότητε, να είναι δημιουργικοί, να μπορούν να δείξουν ηγετικό χαρακτήρα, να μπορούν να δουλέψουν σε μια ομάδα έτσι ώστε να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο υποστηρίζει τη δημιουργικότητα στην Ιλλανδία εμείς έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία μεταρρύθμισης τη ε, δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να απομακρυνθούμε από την ε, αυστηρή ε, εκπαίδευση την οποία ακολουθούσαμε τόσα χρόνια. Τώρα προσπαθούμε να εμφυσίσουμε στους νέους την αγάπη για την εκπαίδευση και τη θέληση των ιδίων να μορφωθούν και να εκπαιδευτούν. Τώρα, το θέμα των πανεπιστημίων. Εγώ προσπαθώ συχνά να ενισχύσω διεθνεί φοιτητέ, φοιτητέ αλλοδαπού να έρθουν να σπουδάσουν στην ε, Ιρλανδία. Και πολύ συχνά το θέμα της κατάταξης των ε, πανεπιστημίων ε, μπαίνει στη συζήτηση. Πρέπει βεβαίω να δούμε για και το θέμα του κατά πόσο είναι δίκαια αυτά τα συστήματα, γιατί πολλέ φορέ επικεντρώνονται μόνο σε έναν κλάδο των πανεπιστημίων και δεν βλέπουν ε, άλλου, όπω α πούμε πόσο ε, συμμετοχικά είναι αυτά τα, αυτά τα πανεπιστήμια, πόσο ενισχύουν τα παιδιά που είναι από ε, μειονεκτούσε οικογένειε να έρθουν να σπουδάσουν. Θα πρέπει λοιπόν όντω να μπορούμε και εμεί από μόνοι μα να ενισχύσουμε, να αξιολογήσουμε συγγνώμη, τους, ε, τα πανεπιστήμια μα. Τώρα, το να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο τη ε, εγκατάλειψη των ε, ε, σχολείων από του μαθητέ είναι πολύ σχηδέ θέμα, είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Πρέπει να το δούμε από την αρχή, από, την, από τον υπηαγωγείο μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε ένα επίπεδο ισότητας σε όλο το, σε όλο το φάσμα. Κυρίως πρέπει να δούμε την, ε, προ, την ε, έγκαιρη μάλλον παρέμβαση, να δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι μαθητές που ε, κινδυνεύουν να φύγουν ή που έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να φύγουν από το σχολείο να τον καταλήψουν και να παρέμβουμε τότε, αντί να παρέμβουμε αφού το έχουν καταλήψει. Για τη διαβίου μάθηση και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, αυτό που θα συζητήσουμε κύριε Κέλλη είναι ο ρόλος των επαγγελματιών εκπαιδευτών των καθηγητών. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι ε, καθηγητές έχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται καθημερινά ε, για να μπορούν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που γίνονται στον κόσμο. Αυτοί λοιπόν που εκπαιδεύουν τους καθηγητές έχουν ζωτικό ρόλο να παίξουν σε όλη αυτή τη διαδικασία και η διάσκεψη το Φεβρουάριο ακριβώς θα συμβάλλει στην εκπόνηση συμπερασμάτων του Συμβουλίου που θα υποστηρίζουν την συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα αυτό. Και αυτά ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθούν το Μάιο, οπότε θα δείτε κάποια πρόοδο, θα υπάρξει πρόοδο σε αυτό. Η κυρία Κάμερβερτ, δεν ξέρω να το είπα σωστά το όνομά σα, μίλησε για την ενεργεία των νέων και την άτυπη εκπαίδευση. Να πω ένα πράγμα εδώ για την διαβίωμα, γενικώ. Υπάρχει ίσω η προσδοκία, κυρίως για τον ιδιωτικό τομέα, ότι αυτό είναι ο ρόλος του κράτους. Εγώ θα έλεγα ότι και ο κλάδο είναι καταναλωτή των, ταλέντων, αλλά πρέπει και να συμβάλλει στην ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων που θέλει μετά να χρησιμοποιήσει. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι ακριβώς που θα απασχοληθούν σε διάφορες εταιρείε ανά την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και οικονομική ενίσχυση, και στην, Ευρω... και στην Ιρλανδία κάποιε από τι ε, επιχειρήσει αυτέ συμβάλλουν οικονομικά. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν και δυνατότητε μαθητεία σε κάποιε τέτοιε εταιρείε για του ε, φοιτητέ. Αν θέλουν λοιπόν να παίξουν το ρόλο του στην διαβίου θα πρέπει να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, κυρία Κάμερμπερτ, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η όλη η διαδικασία τη άτυπη ε, εκπαίδευση. Πολλέ φορέ δεν αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι στου φοιτητέ για το τι μπορούν τελικά να πετύχουν. Στην Ιρλανδία έχουμε ένα, είχαμε έναν ε, νέο, 17 χρονών, έναν κύριο James Welton από το Cork, ο οποίος είδε, για τον οποίο υπήρχε ένα κενό στην εκπαίδευση για, την, για τον προγραμματισμό των ε, ε, υπολογιστών. με αυτό ασχολείται ο συγκεκριμένος νέος Προφανώ οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν πολλά, κάθε μέρα όλο και περισσότερα για του ε, υπολογιστέ. Ο ίδιο ήταν πολύ παθιασμένο με το τομέα αυτό. Οπότε προσπάθησε να δημιούργησε μάλλον μία, ε, μία λέσχη ε, προγραμματιστών ε, ξεκίνησε από μία και τώρα έχουν γίνει 150 λέσχες στην ε, Ιρλανδία όπου ενθαρρύνουν ε, πολίτες από οι εργαζόμενους στον τομέα του προγραμματισμού να έρθουν στις λέσχες αυτές και να βοηθήσουν να ενθαρρύνουν τους μαθητές. Μάλιστα μια τέτοια λέσχη έγινε και στη Silicon Valley. Υπάρχουν στην, υπάρχουν στην Αυστραλία, υπάρχουν στην Αργεντινή. Υπάρχουν λοιπόν αντίστοιχα παραδείγματα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να γίνει ένα τέτοιο, μια τέτοια ε, εκδήλωση και εδώ στις Βρυξέλλες. Έτσι λοιπόν και οι ίδιοι οι νέοι μπορούν να αντιμετωπίσουν από μόνοι τους τις ε, προκλήσεις. Ε, πολλές φορές τους υποτιμούμε. Ευχαριστώ. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω μιλήσει. Θέλω όμως να πω δύο-τρία πραγματάκια. Κύριε Κάνον. Δεν μιλήσατε καθόλου για το πρόγραμμα. Μιλήσατε για την ε, ε, διαβίου μάθηση. Μόνο η κυρία Φιτζέραλτ ε, ανέφερε το όνομα του, προγράμμου, του προγράμματος. εντάξει, δεν θα το αναφέρω ούτε εγώ. υπάρχουν βεβαίως και σημαντικά θέματα. Είμαι και εγώ της άποψης όπως και οι συνάδελφοι ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ε, θα πρέπει να υποστηρίζει και την επίσημη και την, μη, ε, και την άτυπη εκπαίδευση. πρέπει να ενισχύσουμε τους ε, μακροχρόνια άνεργους να, ε, να λάβουν νέες δεξιότητες, να έχουν νέα πληροφόρηση, αλλά αυτό πρέπει να γίνει στα πλαίσια του προγράμματος που υπάρχει για αυτό το σκοπό. Σας παρακαλώ λοιπόν σε αυτό το τομέα και στην Κορεπέρ ή όπου πάτε, εν πάση περιπτώσει, όπου το συζητήσετε, να φροντίσετε ώστε σε αυτό το κοινωνικό ταμείο για το οποίο λέει η Κομισιόν ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει, να αναφερθεί ρητά αυτό. Αν δεν αναφερθεί ρητά, δεν πρόκειται και να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνέχεια να υπεραμεινόμεθα των πράξεών μας γιατί πάντα μας ρωτούν ναι αλλά δεν γίνεται αυτό στα πλαίσια του Λεωνάρντο είναι δυνατόν να γίνει στα πλαίσια του Λεωνάρντο Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την, μέχρι το τέλο τη εκπαιδευτική λυσίδα. Από εκεί και μετά πρέπει να παρέμβει το κοινωνικό ταμείο. Και αυτό θα ήθελα να σα ζητήσω να προωθήσετε. πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, το είπαν και οι συνάδελφοι και το είπατε κι εσείς, όταν μιλούμε για την εκπαίδευση και την παιδεία. Εγώ θυμώνω πάντα όταν η Κομισιόν ε, λέει ότι για το 2020 χρειαζόμαστε 40% ε, ε, ε, πτυχία πανεπιστημιακά. Αυτά είναι αηδίες. Δείτε πόσοι έχουν πτυχίο στην Ισπανία και δεν έχουν δουλειά. Και χρόνια τώρα. Το θέμα δεν είναι να έχεις πτυχίο, είναι να έχεις μια καλή εκπαίδευση. Και εμείς στην ε, Γερμανία μιλούμε και για ένα θέμα, για, ένα, για μια ισοδυναμία πτυχίου. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα δεν είναι ότι είναι γερμανικό αυτό το σύστημα και γι' αυτό είναι καλό. Είναι καλό γιατί λειτουργεί. Δεν, γιατί δεν είναι δυνατόν αυτό το διπλό σύστημα να εισαχθεί ακριβώς εκεί όπου υπάρχουν και μεγάλες μικρές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να συνεργαστούν με τα πανεπιστήμια και να προετοιμάσουν τους νέους για μια ζωή όπου θα μπορούν να εργάζονται και στην δουλειά τους θα μπορούν να παραμείνουν ε, ή θα μπορούν και να φύγουν ε, αν δεν το θέλουν ε, και θα μπορούν να προχωρήσουν γενικώ. Δεν μπορεί να, αν θέλουν να επιστρέψουν στο πανεπιστήμιο. Αλλά πείτε μου, Ποιο είναι αυτός ο, ε, ο μηχανικός που σας ε, διορθώνει τον ε, καυστήρα όταν χαλάσει ή σας ε, βάζει τα, τα πατώματα. Έχει πτυχίο αυτός που σας βάζει τα πατώματα. Ας δούμε λίγο την πραγματικότητα. Ας δούμε πώς έχει το πράγμα. Α μην χανόμαστε μέσα σε αυτά τα πολλά προγράμματα. Πρέπει να προσπαθήσουμε του νέου να του οδηγήσουμε εκεί ακριβώ που υπάρχουν δυνατότητε εργασία αλλά για την οποία εργασία θα είναι εκπαιδευμένη. Μπορούμε πάντα να μιλούμε για ε, τους ε, πτυχιούχους, τους 40%, 50%, μπορούμε να θέλουμε και 100%. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ήθελα λοιπόν να τα πω αυτά, γιατί είναι θέματα που με απασχολούν. Τα τελευταία χρόνια αυτές τις βέλτιστες πρακτικές που κυκλοφορούν από χώρα σε χώρα δεν τις υιοθετούμε. Είναι λοιπόν ε, σημαντικό για μας στην ε, διάρκεια της Προεδρίας σας να το προωθήσετε αυτό. Όχι γιατί αυτό το θέμα είναι γερμανικό, είναι σύστημα γερμανικό και λειτουργεί, αλλά γιατί είναι λειτουργικό από μόνο το σύστημα, ανεξαρτήτως του ότι είναι γερμανικό. Αυτό ήθελα να πω. Τι άλλο ήθελα να πω. Α, το θέμα με τα κονδύλια. Έπρεπε να σας είχα μαζί μου εχθές στο Bundestag, στην Άνω Βουλή. Ε, η κυρία Μέρκελ λοιπόν έκανε μια πολύ ωραία ομιλία. Επίσης ο κύριος Ολόντ μια εξαιρετική ομιλία και οι δύο μίλησαν για την παιδεία όχι για όλη την ε, ομιλία του, αλλά ένα τρίτο τη ομιλία του είχε να κάνει με την παιδεία, με την εκπαίδευση, με το πόσο σημαντικό είναι. Εγώ χειροκροτούσα συνέχεια, δεν σταμάταγα. Πρέπει λοιπόν να τα πάρουμε σοβαρά αυτά που λένε και στην επόμενη συνεδρίαση πρέπει να πείτε ότι ξέρουμε ότι στις, ε, στους εορτασμούς ε, με την Μέρκελ και τον Ολόντ αναφέρθηκε το θέμα της παιδείας και εκεί πρέπει να πάνε τα κονδύλια. Δεν σας λέω ψέματα, υπάρχουν και γραπτό όλα αυτά που σας λέω. Πρέπει πραγματικά να το προωθήσουμε αυτό. Ξέρουμε ότι ε, μόνο ένα μικρό κομματάκι των κονδυλίων πάει στην εκπαίδευση και στην παιδεία. Αλλά πραγματικά δεν είναι τίποτα. Είναι... Ε, αν μειωθούν ακόμα ε, περισσότερο τα κονδύλια, δεν θα αλλάξει τίποτα για τα υπόλοιπα προγράμματα, αλλά για μας θα είναι σημαντικό. Σας παρακαλώ λοιπόν να φροντίσετε ώστε το Φλεβάρι να ενισχυθεί και το, να, να ε, τονιστεί το θέμα αυτό και να ε, ζητήσετε ο προπολογισμό να παραμείνει ο ίδιος τουλάχιστον, αν όχι να αυξηθεί. Δεν, δεν είναι υπερβολικό αυτό που σας λέω. Πρέπει να έχουμε τα χρήματα αυτά, γιατί αλλιώς δεν, δεν, ε, δεν, θα, δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα και δεν θα παίρνουμε εμεί τα λεφτά. Οι νέοι μας τα παίρνουμε. Μακάρι λοιπόν τέλος του επόμενου μήνα να έχουμε τα κονδύλια έτσι ώστε και γρήγορα μετά από αυτό να μπορέσουμε να περάσουμε στη διαδικασία συναπόφασης και να λύσουμε και τα υπόλοιπα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε ε, Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους για την πολύ καλή συζήτηση που κάναμε και κλείνουμε την συνεδρίαση μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.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 and look at the lady of the Corepair. She, was, she, was, she was giving you the idea, right? I, I know. I thank very much the lady from the Corepair. Ευχαριστώ. την κυρία από την Κορεπέρ για τις συμβουλές που δώσε στον κύριο Κένον. Λοιπόν, όποιος θέλει να μείνει μπορεί να μείνει, όποιος δεν θέλει πρέπει να περάσει. Εκτός εθούσης, είμαστε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, προϋπολογισμός, ε, απαλλαγή, γενικός προϋπολογισμός, η κυρία Λόκεγκαρντ, ο, ο ε, κύριος Λόκεγκαρντ έχει το λόγο, συγγνώμη. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Δεν θα κρατήσουμε τη συζήτηση για πολύ διάστημα, θα είμαι σύντομος. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πρόβλημα. Δεν είναι πολύ αμφιλεγόμενο το θέμα φέτος. Το δικό μας κομμάτι του προϋπολογισμού τουλάχιστον δεν είχε προβλήματα και είχαμε και κάποιες βελτιώσεις, θα τις πω εντάχει. Δεν ξέρω αν έχετε το έγγραφο μαζί σας. Εμείς προτείνουμε, εγώ προτείνω πέντε σημεία. Τα τρία τεχνικού χαρακτήρα. Κάποιες λεπτομέρειες που ήταν κομμάτι των εκθέσεων μέχρι τώρα. Μίλαμε για βελτιώσεις στην υπηρεσία, στην εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαίδευσης και κατάρτισης γρήγορες πληρωμές ε, βασικά και νομίζω ότι μας χαροποιεί το ότι η υπηρεσία στον τομέα αυτό δουλεύει καλά. Βελτιώσεις και εδώ. Κατόπιν μας ανησυχούν τα λάθη στις συναλλαγές ε, στην υπηρεσία διαβίου εκπαίδευσης. Κάποια από την έλλειψη επαιτούμενων δικαιολογητικών από πλευρά των δικαιούχων και μη τήρηση των κανόνων ε, ε, ε, ανάληψης ευθύνης. Είναι το μόνο που μας ανησυχεί. Τέταρτο σημείο. Καλωσορίζουμε τις βελτιώσεις στα εθνικά συστήματα ελέγχου των εθνικών υπηρεσιών και ένα πέμπτο σημείο που με ικανοποιεί ιδίως είναι ότι τα πιλωτικά σχέδια ξεκίνησαν εκ νέου μετά τη διακοπή του 2010. Φαίνεται ότι έκτοτε η Επιτροπή το ξανασκέφτηκε και έχουμε ένα συμπληρωματικά να σας πω ότι διάβασα διαβάζω πιο σωστά τη νέα έκθεση της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου για την ε, ελευθερία των μέσων. Στη σελίδα 29 υπάρχουν 30 συστάσεις. Η, 14, η 14η αφορά το θέμα αυτό, την ανάγκη υποστήριξης και δημιουργίας νέων τρόπων χρηματοδότησης ε, διασυνοριακής δημοσιογραφίας Μα υποστηρίζει λοιπόν ε, αυτή η ομάδα υψηλού επισπέδου που νομίζω ότι μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι το έργο είναι πάντα ζωντανό. Αυτά είναι τα τέσσερα, τα πέντε βασικά σημεία. Περιμένω το σχόλιά σα. Κύριε Κέλλη. Ναι. Εκ μέρου του κυρίου Μπέλετ ε, θα σχολιάσω. Δεν μπορούσε να είναι εδώ. Ήταν εδώ το πρωί για την πρώτη, ε, για την ανταλλαγή απόψεων την έκθεσή του, όμως ε, έχει πάει σε μια συνάντηση της αντιπροσωπείας του. Το ΕΛΚ θα ήθελε να τονίσει ότι υποστηρίζουμε πλήρως την έκθεση του εισηγητή. Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για την εξαιρετική του δουλειά. Είμαστε ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι δεν ε, ανοιχνεύτηκαν σφάλματα την οικονομική χρήση 2011 σε σχέση ε, με τις αρμοδιότητες αυτές ε, ε, σε σχέση δηλαδή με την υπηρεσία για τον οπτικοκουστικό τομέα, τον πολιτισμό και τα λοιπά Δεν υπήρξαν ε, παράπονα από τους εμπλεκόμενους φορείς, ε, όμως επιμένουμε ότι πρέπει να δοθεί ε, περισσότερες, περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στους δικαιούχους σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους και θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι πάντοτε υποστηρίξαμε την συμμετοχή στον αθλητισμό Έχουμε βέβαια του περιορισμού του τρέχοντος προπολογισμού, θέλουμε όμως μεγαλύτερη φιλοδοξία από την Επιτροπή. Έδωσε το Κοινοβούλιο πολλές ε, συστάσεις στην ε, Επιτροπή για προπαρασκευαστικές εργασίες. Το 2013 θα είναι πολύ κρίσιμο έτος για την Επιτροπή για να δείξει ότι είναι ικανή για πρώτη φορά να ε, λειτουργήσει ένα πραγματικό πρόγραμμα αθλητισμού που θα αρχίσει το 2014. Εμείς περιμένουμε βεβαίως ε, με αγωνία να ολοκληρωθεί αυτό σε ε, στενή συνεργασία με την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ στον, τον Μόρτεν Λόκεγκαρτ. Χαίρομαι που ακούω ότι δεν υπάρχουν σοβαρά σφάλματα γιατί τα τελευταία χρόνια είναι πολύ υψηλό το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού στα προγράμματά μας. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε και μεγαλύτερο προϋπολογισμό, γιατί δεν είναι ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε, συνήθω το ανάποδο συμβαίνει. Υπάρχουν πολύ περισσότερες ανάγκες από αυτά που ε, ο προπολογισμό μας μπορεί να καλύψει. Είναι όμως πολύ καλό να ξέρει κανείς ότι η εφαρμογή λειτουργεί και ότι δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς για απάτες, ε, ε, ή μεγάλα προβλήματα στο σύστημα. Θα ήθελα απλώ ένα πράγμα να, τον, να τονίσω, το οποίο είπε και εσύ, Μόρτεν, το διασυνοριακο διασυνοριακή δημοσιογραφία. Ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να το αναγνωρίσουμε και θα ήθελα πραγματικά να το ενθαρρύνω. Χαίρομαι που στο σημείο 1 αναφέρεται Ε, αναφέρονται κάποια αιτήματα που γίνονται πάντα. Ίσως ε, πολλά μπορεί να τα, μπορούμε να τα δούμε και όσο καταποκοπή ποσά. Ε, τα λάθη τώρα που αναφέρθηκαν νομίζω ότι προέκυψαν για το ότι ζητήθηκαν ας πούμε 5.000 ή 20.000 ευρώ σε διοικητικό επίπεδο. Δεν είναι δηλαδή απάτη. Ε, την απάτη τη βρίσκουμε στα 2 εκατομμύρια ή στα 200 χιλιάρικα, όχι, ή στα 200 εκατομμύρια, όχι τώρα στα 5.000 ευρώ. Ε, νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Κομισιόν. Ποιο θα μιλήσει εκ μέρου τη Κομισιόν, ποιο θέλει να μιλήσει εκ μέρου τη Κομισιόν, παρακαλώ. Um, Martine είμαι εδώ για την Γενική Διευθυνσία που είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη από την υποστήριξη που δίνεται στις βελτιώσεις ε, του κειμένου που θέσαμε για να μειωθούν τα ποσοστά σφάλματος. Νομίζω ότι σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης δουλειάς στον τομέα αυτό και θέλουμε και εμείς να το υπογραμμίσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι όπως είπατε και εσείς η υλοποίηση των προγραμμάτων σε επίπεδα εκτέλεσης είναι καλή και η αλυσίδα ελέγχου λειτουργεί καλά. Αυτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν. 29 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες σας. Πάμε στο σημείο 11. Έχουμε ένα πρόβλημα με τους ε, συντονιστές, με τα όσα διαμήθησαν στη συνεδρίασή τους. Το θέμα των μελετών που πρέπει να ετοιμαστούν για μας αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση, που θα γίνει το Φλεβάρι. Αλλά αυτό δεν γίνεται, γιατί αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τούτε τι μελέτε πρέπει να περιμένουμε, πρέπει να περιμένουν και να μην κάνουν τίποτα ε, μέχρι το Φλεβάρι. Οπότε, μάλλον αυτό έγινε γιατί ο κύριο Ταβάρη και ο κύριο Τάκουλα ε, είχαν διαφορετική αντίληψη για το τι θα πρέπει να μελετηθεί. Εγώ δεν έχω αντίρρηση με αυτό, αλλά αυτό που έχουμε στα χέρια μας σημαίνει είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε μέσα στην, ε, στην, ε, στο χρόνο. συνήθως ε, εγκρίνουμε τα όσα λένε οι συντονιστές και δεν το πολύ θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε ε, εγώ να δώσω την ε, ευχή μου, ας πούμε, στους, σε όσους έχουν αναλάβει έκθεση, να ξεκινήσουν και μόλις έχουν ολοκληρώσει μια από τις εκθέσεις, να δούνε και τις νέες προτάσεις του Ταβάρες και του Τάκουλα. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι ένας ε, κανονικός, ικανός τρόπος για να λειτουργήσουμε. Ε, καταλάβατε τι εννοώ. Υπάρχουν πολλές μελέτες. Μπορείτε να μας πείτε ποιες μελέτες, ποιες εκθέσεις θα κάνετε. Το έχουμε όλοι, αλλά καλό είναι να μας το πείτε κιόλα. Πείτε μας. Ευχαριστώ. Η πρώτη στηρίζεται στο πρόγραμμα εργασία τη Επιτροπή. Η διεθνοποίηση τη διεθνού της, η διεθνοποίηση της ε, ε, ε, εκπαίδευσης. Προ, της, της διεπαφής, η ιστορική μνήμη της εκπαίδευσης στην Ευρώπη, η ανακοίνωση για την Ευρώπη του και τους πολίτες και η διδασκαλία των εκπαιδευτικών. Μια παρατήρηση. Σε μία από τις δικές μου προτάσεις ε, αναφερθήκατε που είπε το, στους συντονιστές ο κ. Στάκουλα. Να προσθέσω ωστόσο, αν είναι για το θέμα αυτό, Τι είχατε προτείνει λέει η πρόεδρος. Γίνεται μια σημαντική συζήτηση στη Σκανδιναβία και αλλού για το μέλλον της αγοράς βιβλίου. Προσπάθησα να βρω αν υπάρχουν πρόσφατες μελέτες, αν είναι στη μέση διάταξη της Επιτροπής μας, από ό,τι φαίνεται όχι. Είναι σημαντικό θέμα. Μιλάμε για το μέλλον του βιβλίου που απειλείται από την απελευθέρωση. Τουλάχιστον αυτό λένε οι βιβλιοπόλες. Μπορούμε να κάνουμε μια μελέτη για το πώς τα κρατημέλη αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό. Γιατί το αντιμετωπίζουν με τελείως διαφορετικό τρόπο και χρειαζόμαστε κάποια στοιχεία. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ πράγμα, αλλά κάτι, της μια μελετούλα. Μπορεί να υπάρχει παρανόηση ή εγώ τα μπλέξα. Όταν μιλήσαμε στους συντονιστές σήμερα, πολλοί συνάδελφοι θεωρούσαν ότι το θέμα ήταν προτάσεις για τις μελέτες στις οποίες θα έπρεπε να προχωρήσουμε. Αυτή ήταν η άποψη των φιλελευθέρων και της δικής μου ομάδας. Προφανώς αυτό δεν ήταν η κατάσταση, αλλά εξού και η σύγχυση. Η εντύπωσή μας είναι να υποβάλουμε, να παρουσιάσουμε νέες μελέτες, όχι να δούμε ποιες μελέτες προχωρούν αυτή τη στιγμή. Θα στείλουμε μια επιστολή στους συντονιστές. Νομίζω συνεχίστε τις, δουλειά, τις μελέτες που κάνετε. Μόλις τελειώσετε κάτι, ξεκινήστε με κάτι που προτάθηκε σήμερα. Αυτό που λέει ο κύριος Λόκεγκατ δεν είναι δικό μας θέμα. Εγώ δεν πρόκειται να παραιτηθώ, γιατί είναι θέμα που ανήκει στην ΕΚΟΝ. Δεν είναι δικό μας θέμα. Η Επιτροπή δεν έχει, να κάνει, δεν έχει σχέση με εμά. Είναι εμέσω συνδεδεμένη με τη δική μα την ε, Επιτροπή και, την, ε, και τον πολιτισμό. Ναι, αλλά αυτό είναι θέμα πολιτισμού. Όλες αυτές οι πολιτικές θα έχουν επίπτωση στη συζήτηση για την ε, πολιτιστική διαφοροποίηση. Και αυτά είναι και τα επιχειρήματα των εκδοτών, των βιβλιοπολών, ότι δηλαδή δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά λένε ότι θα οδηγήσει σε λιγότερους τίτλους, λιγότερα βιβλία και αυτό θα ε, πειράσει αυτό που θέλουμε να διαφυλάξουμε, την πολιτιστική ε, διαφοροποίηση. Νομίζω δηλαδή ότι είναι αμυγός πολιτιστικό θέμα. Εντάξει, αλλά εγώ είμαι πολλά χρόνια εδώ και ξέρω ότι ε, έχουμε έκθεση για αυτό το θέμα ότι ε, η, αυτό το θέμα έχει γίνει αποδεκτό και δεν ε, έχει αλλάξει. Αυτό, αυτό που είπες δεν έχει γίνει. Ούτε λιγότερα ε, βιβλία εκδόθηκαν, ούτε λιγότερα βιβλία τυπώθηκαν, ούτε τίποτα. Λοιπόν, είναι θέμα στατιστικής, αν θέλεις. Οπότε μπορείτε να το κάνετε έτσι παράλληλα. Εντάξει, ωραία. Το κλείσαμε κι αυτό. Το πρόβλημα τώρα του Ταβάρες Ήθελε κάτι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πού είναι, βρέστο μου. Ίσως να μπορούσαμε το θέμα αυτό του Ταβάρες. Μπορείτε να με ακούσετε λίγο εκεί πίσω. Σε παρακαλώ. Ο κύριος Ταβάρες μίλησε για ένα θέμα σχετικό με την ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κάτι με τα σχολεία, δεν θυμάμαι πόσα Πώ μπορούν τα, ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να συνεργαστούν και μια, να κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας γι' αυτό, να γίνει μια μελέτη γι' αυτό. Ωραία. Εντάξει, το δυναμικό των ε, ε, πανεπιστημίων. Εσείς θα κάνετε μια έκθεση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα την κάνετε. Δεν θα την κάνετε. Ναι, ναι. Μία μελέτη μια μελέτη αφορά τη διεθνοποίηση τη ανώτερη εκπαίδευση, μια βασική πρόκληση και που είναι κομμάτι του προγράμματο Εργασία Επιτροπή για το 2013. Είπαμε ότι θα ήταν σκόπιμο να σταθούμε εκεί για να κάνουμε μια μελέτη για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και να είμαστε και επαρκώς ε, εξειδικευμένοι για να έχει μελέτη ουσία. on the education, on the higher education system and on the university situation. Θα μπορούσε να μιλήσει ο κύριος Ταβάρης μαζί σας και να διευρύνουμε το θέμα. Ναι, πολύ ωραία ιδέα. Να το πείτε εσείς τον κύριο Ταβάρες. Ωραία. Και μετά να δώσουμε όλη τη θεματική στους υπεύθυνους των μελετών. Θέλετε το λόγο? Βέβαια. Έχουμε και άλλη πρόταση μελέτης για τη σύνδεση της εκπαίδευσης στην ανώτερη εκπαίδευση με την καινοτομία, που εν μέρη μπαίνει στο ίδιο θέμα. Δίκιο έχετε. αυτό που κάνουμε, όλο ό,τι κάνουμε για τα πανεπιστήμια συνδέονται μεταξύ τους. Δείτε τι θέλει ο Ταβάρες και εντάξτε το σε αυτά που κάνετε ήδη. Να μιλήσουμε. Πολύ ωραία. Λύσαμε το πρόβλημα. Όλοι είναι ευτυχείς, πράσινοι, φιλελεύθεροι και λοιποί. Κάντε λοιπόν μελέτες, διάφορα, όχι. 20 Φεβρουαρίου επόμενη συνάντηση. 21. 21